σας καλωσορίζω στην πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής μας μετά τις καλοκαιρινές διακοπές. Δυστυχώς ε, η Πέτρα δεν μπορεί να είναι εδώ, έτσι λοιπόν θα προεδρεύσω εγώ. Το πρώτο σημείο στην ημερήσια διάταξη είναι η έγκριση της ημερήσιας διάταξης, αν δεν έχετε αντιρρήσεις. Θα πρότεινα να αλλάξουμε τη σειρά των δύο ψηφοφοριών γιατί ο κύριος Λόκεργκαρτ ε, θα καθυστερήσει, θα έρθει σε λίγα λεπτά γιατί έχει εγκλωβιστεί σε συμφόρηση. Αν δεν έχετε λοιπόν αντίρρηση να αλλάξουμε τη σειρά των δύο σημείων για ψηφοφορία. Δεν βλέπω αντιρρήσει. Το δεύτερο σημείο είναι η έγκριση των πρακτικών των συνεδριάσεων της 18 η 19 η ιουνιου 2018 Έχουν ε, κατατεθεί τα πρακτικά. Έχετε παρατηρήσει σχόλια. Αν όχι, προτείνω να θεωρήσουμε ότι εγκρίνονται τα πρακτικά. Αν ε, δεν γίνουν μέχρι το τέλος συνεδρίσεις κάποιες παρατηρήσεις. Προχωράμε στις ανακοινώσεις της Προέδρου. Καταρχήν για την ε, διερμηνία. Έχουμε διερμηνία σήμερα σε γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, αγγλικά, ελληνικά, ισπανικά, τσεχικά, εσθονικά, ουγγρικά, πολωνικά, βουλγαρικά και ρουμανικά. Ευχαριστώ και τους διερμηνείς και να σας υπενθυμίσω ότι η συνεδρίασή μας αναμεταδίδεται ζωντανά στο διαδίκτυο. Μπορείτε να την παρακολουθήσετε στο ιστοσελίδα του Κοινοβουλίου. Το επόμενο θέμα στην ημερησία διάταξη είναι οι ψηφοφορίες. Ετοιμαστείτε παρακαλώ, ετοιμάστε τις κάρτες σας, θα ξεκινήσουμε με μια πρόταση ψηφίσματος προώθηση της αυτόματης αμοιβαίας αναγνώρισης διπλωμάτων. Και πριν να περάσουμε στη ψηφοφορία, να έχετε κατά νου ότι έχουν κατατεθεί από τους φιλελευθέρους δύο προφορικές τροπολογίες. Να ξεκινήσουμε λοιπόν με την ψηφοφορία. Λοιπόν, πρόθεση της αυτόματης αμοιβαίας αναγνώρισης των διπλωμάτων και των αποτελεσμάτων των περιόδων εκμάθησης στο εξωτερικό. Λοιπόν, συμβαστική τέσσερα υπέρ, κατά. Αποχές, εγκρίνεται. Να περάσουμε στη συμβαστική 5. Υπέρ. Κατά. Εποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 22. Υπέρ. Κατά. εποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 24. Υπέρ. Κατά. εποχές εγκρίνεται. 23. Συγγνώμη. 37. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 6. Υπέρ. Παρακαλώ. Να ελέγξουμε την 37. Ε, να ελέγξουμε λοιπόν την τροπολογία 37. The vote is closed. Λήξη. Εγκρίνεται. Περνάμε στην συμβιβαστική 6 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 31 υπέρ. Mm. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 34 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 35 υπέρ με την προφορική τροπολογία 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 5 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 13 υπέρ. Κατά. Αποχές συγκρίνεται. 14 υπέρ. Κατά. Αποχές συγκρίνεται. 15 υπέρ. Κατά. Αποχές συγκρίνεται, 16 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 1. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 3 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 4 με την προφορική τροπολογία 1 υπέρ. Κατά εποχέ, συγκρίνεται. Περνάμε στην τελική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισατε όλοι. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια. The result is 19 Uh, 19 υπέρ, κανένα κατά και μία αποχή. Πολύ καλό το αποτέλεσμα. Mm-hmm. Then we have come to Περνάμε τώρα στη δεύτερη ψηφοφορία στο σχέδιο γνωμοδότησης του κυρίου Λόκιγκαρτ. Νομίζω έχει καταφτάσει. Έχετε το λόγο. I think we just move on. Μπορούμε να προχωρήσουμε νομίζω. Πολύ ωραία. Α περάσουμε στην ψηφοφορία. Τροπολογία 1, υπέρ. Κατά. Αποχές. εγκρίνεται. 3, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 4 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 5 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 6 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 7 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 9 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται. 10 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται. 12 υπέρ κατά εποχές απορρίπτεται. 11 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται 14 υπέρ κατά εποχές απορρίπτεται 13 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 16 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 17 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 19 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 20 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 21 βερ, κατά εποχές εγκρίνεται. Περνάμε στην τελική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 17 υπέρ, 5 κατά. Καμία αποχή. Συγχαρητήρια στον εισηγητή. Mr. Lockegaard. Κύριε Λόκιγκαρτ, θέλατε το λόγο. Μόνο για να ευχαριστήσω όλους τους συμμετέχοντες. Οι συζητήσεις και οι διαπραγματεύσεις ήταν πάρα πολύ καλές. Απέδωσαν καρπούς. Οι τροπολογίε είναι καλές και νομίζω πως έχουμε καταφέρει ε, να βελτιώσουμε το αποτέλεσμα. Γι' αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συμμετέχοντε τη Γραμματεία και τους βοηθούς. Σας ευχαριστώ πολύ για τη δουλειά σας. Έπειτα, η πρόταση ψηφίσματος ψηφίστηκε στην αρχή, ε, θα ήθελα να πω ότι πέρα από τις προφορικές τροπολογίες, τα μέλη θα ασκήσουν πίεση στις δικές τους πολιτικές ομάδες και θα το συζητήσουν έτσι ώστε να συζητηθεί το θέμα στην πρώτη ολομέλεια του Οκτωβρίου. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να παρακαλέσω τους προέδρους των πολιτικών ομάδων να το πράξουν. Συνεχίζουμε όμως με το επόμενο σημείο, σημείο 6 στην ημερήσια διάταξη. Μία έκθεση πρωτοβουλίας για την Ευρωπαϊκή Ατζέντα για τον Πολιτισμό. Η συγητής είναι ο κύριος Γραμματικάκης από την ομάδα S&D. Προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών είναι η 12η Σεπτεμβρίου, 12 η ώρα το μεσημέρι και στις 20 Νοεμβρίου θα συζητηθεί το θέμα στην Επιτροπή μας έτσι ώστε το Δεκέμβριο να ε, συζητηθεί στην Ολομέλεια. Όπως γνωρίζετε, πριν το καλοκαίρι έγινε μια δημόσια ακρόαση για την Ευρωπαϊκή Ατζέντα για τον πολιτισμό που ακούσαμε τις απόψεις των εμπειρογνωμόνων. Ελπίζω η συνεισφορά να ήταν σημαντική σε αυτήν την έκθεση πρωτοβουλίας την οποία για πρώτη φορά θα συζητήσουμε στην Επιτροπή μας. Θα ήθελα λοιπόν, χωρίς ε, περαιτέρω καθυστερήσεις, να δώσω το λόγο στον ε, ε, εισηγητή, ο οποίος από τον Ιούλιο μέχρι τώρα έχει εργαστεί πάρα πολύ σκληρά. Έχετε πέντε λεπτά χρόνο, κύριε Γραμματικάκη. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Η νέα Ευρωπαϊκή Ατζέντα για τον πολιτισμό αποτελεί πράγματι μια ιστορική ευκαιρία διότι μας δίδει τη δυνατότητα να διαμορφώσουμε μια συντονισμένη ευρωπαϊκή πολιτική για τον πολιτισμό και τις εκφράσεις του. Θα ήθελα λοιπόν ως εισηγητής να χαιρετήσω την πρόταση της Επιτροπής που έρχεται μάλιστα σε μια σημαντική χρονική στιγμή καθώς φέτος διανύουμε το Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Ο θεσμός αυτός υπενθύμησε και στους πιο αδιάφορους ότι ο πολιτισμός είναι ένας σπουδαίος, ίσως ο πιο σπουδαίο συνδετικός κρίκος για τους λαούς της Ευρώπης. Αξίζει μάλιστα να τονιστεί ότι η αξία του πολιτισμού δεν είναι μόνο άειλη. Το αντίθετο μάλιστα, η προστιθέμενη αξία των δημιουργικών τομέων ανέρχεται περίπου σε 509 δισεκατομμύρια ευρώ, πράγμα που ισοδυναμεί ούτε λίγο ούτε πολύ με το 5,3% του ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η νέα ατζέντα για τον πολιτισμό μπορεί ωστόσο να επιτύχει τους φιλόδοξους στόχους που θέτει μόνο εάν συνοδεύεται από μια σημαντική αύξηση των πόρων της. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη που ανώ απέκτησε μεγάλη απήχηση δεν έχει την ανάλογη χρηματοδότηση. Αρκεί να σημειωθεί ότι η χρηματοδότηση αυτή αντιπροσωπεύει μόλις το 0,15 του συνολικού προϋπολογισμού ενώ μόνο το 1 τρίτο του ποσού αυτού προορίζεται για τον πολιτισμό. Με συνέπεια ένα απογοητευτικό 16% των προτάσεων μόνον να δέχεται την οικονομική στήριξη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι λοιπόν ένα πρώτο θετικό βήμα η πρόταση της Επιτροπής για την αύξηση της χρηματοδότησης του προγράμματος. Δεν επαρκεί όμως. Στην έκθεσή μου ζητώ το διπλασιασμό του προϋπολογισμού μετά το 2020. Είναι καιρός αγαπητοί συνάδελφοι, τα μεγάλα λόγια για την αξία του πολιτισμού που ακούγονται συχνά από ηγέτες της Ευρώπης αλλά και την ίδια την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να έχουν και ένα ορατό αντίκρισμα. Παράλληλα, η ανάγκη να ανταποκριθούμε σε απρόβλεπτες προκλήσεις δεν πρέπει να οδηγεί στην ανακατονομή των πόρων του, όπως είναι η συνήθις πρακτική. Αξίζει επίση να αναφερθεί ότι η αποτελεσματική στήριξη των καλλιτεχνικών και δημιουργικών τομέων απαιτεί μια βαθύτερη γνώση της λειτουργία τους. Αυτό συνεπάγεται την ύπαρξη στοιχείων που απουσιάζουν ή είναι συχνά ανεπαρκή. Καλό λοιπόν την Επιτροπή και τα κράτη-μέλη να αναπτύξουν νέε προσεγγίσεις στη συλλογή δεδομένων. Είναι επίση ιδιαίτερα σημαντικό ότι η νέα ατζέντα θα δώσει έμφαση στην κοινωνική διάσταση του πολιτισμού. Ο πολιτισμός αποτελεί δημόσιο αγαθό και η πρόσβαση των πολιτών στις εκφράσεις του πρέπει να ενθαρρύνεται. Θα ήταν χρήσιμο, για παράδειγμα, αν τα κράτη-μέλη φρόντιζαν ώστε οι τέχνες και η δημιουργική σκέψη να συμπεριλαμβάνονται σε όλα τα στάδια εκπαίδευσης και κατάρτισης. Πρέπει επίσης να αυξηθεί η διασπορά των ευρωπαϊκών έργων τέχνης, καθώς και η κινητικότητα των καλλιτεχνών η ειδική δράση που προτείνει η Επιτροπή αποτελεί μια σημαντική πρωτοβουλία. Είναι όμως ανάγκη όπως πάντα να συνοδεύεται από επαρκή χρηματοδότηση αλλά και απλουστευμένους κανόνες προκειμένου να αποφευθούν η διπλή φορολόγηση και οι δυσκολίες της θεωρήσης βίζας. Στην έκθεσή μου ζητώ επίσης τη δημιουργία μιας ενιαίας ψηφιακής πύλης που θα περιέχει πληροφορίες σχετικά με όλα τα διαθέσιμα προγράμματα φιλοξενίας των καλλιτεχνών. Εισηγούμε ακόμα τη δημιουργία μιας ενιαίας φιλική προς το χρήστη πλατφόρμας που θα περιέχει πληροφορίες σχετικά με όλα τα διαθέσιμα προγράμματα επιχορηγήσεων. Είναι βέβαια γεγονός αυτονόητο ότι δεν μπορεί να υπάρξει τέχνη χωρίς τους καλλιτέχνες, ούτε πολιτιστική δημιουργία χωρίς τους δημιουργούς της. Τα κράτη-μέλη πρέπει συνεπώς να δεσμευτούν όσον αφορά τη βελτίωση των κοινωνικών και οικονομικών συνθηκών των καλλιτεχνών. Α σημειωθεί ότι η έλευση της ψηφιακής επανάστασης έχει δυσχεράνει ακόμα περισσότερο τη θέση των καλλιτεχνών και υπό το πρόσχημα της ευρύτερης πρόσβασης τα έργα όπως γνωρίζετε καταλήγουν συχνά να γίνονται αντικείμενα υποκλοπής και παράνομης εκμετάλλευσης. Παράλληλα όμως η ψηφιακή επανάσταση παρουσιάζει και σημαντικές ευκαιρίες για τη διάδοση του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Γι' αυτό και στην έκθεσή μου ζητώ την ανάπτυξη μιας ψηφιακής πλατφόρμας που θα παρέχει πρόσβαση σε επιλεγμένες, για παράδειγμα, ταινίες του ευρωπαϊκού κινηματογράφου, ενώ θα αποζημιώνει φυσικά τους δημιουργούς για το έργο τους. Θα ήθελα επίσης να χαιρετήσω το γεγονός ότι η πρόταση της Επιτροπής δίδει έμφαση στους επιμέρους καλλιτεχνικούς τομείς. Ιδιαίτερα επισημαίνω την πρωτοβουλία Music Moves Europe, η οποία ευελπιστώ ότι θα ενσωματωθεί στο πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη και βέβαια με σταθερή χρηματοδότηση. Είναι περιττό να πω ότι η μουσική είναι μια πραγματικά διεθνής γλώσσα που ανώνει λαούς και πολιτισμούς. Τελειώνοντας, θα ήθελα να σταθώ στην εξωτερική διάσταση της ατζέντα. Είναι απαραίτητη νομίζω η άμεση εφαρμογή της στρατηγικής για διεθνείς πολιτιστικές σχέσεις, καθώς ο πολιτισμός αποτελεί, το επαναλαμβάνω, το δυνατότερο όπλο της Ευρώπης. Εάν λοιπόν η πολιτιστική αυτή διπλωματία αποκτήσει συνέπεια και όραμα, μεγάλα θα είναι τα ευεργετήματα της Ευρώπης. Θα ισχυροποιήσει τις φιλίες και τις διεθνείς της σχέσεις, αλλά θα κερδίσει νέους και πολύτιμους φίλους, ενώ έχω την ελπίδα ότι θα δημιουργήσει νέες ευκαιρίες στους ταλαντούχους Ευρωπαίους δημιουργούς. Με αυτή την αισιόδοξη προοπτική σας ευχαριστώ όλους για την προσοχή σας και περιμένω βέβαια με ενδιαφέρον τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Γραμματικάκη. Τώρα το λόγο θα πάρουν οι σκιώδεις εισηγητές. Ποιος θα ήθελε να προσθέσει κάτι στο θέμα αυτό. Ένα σκιώδης εισηγητής έχει δηλώσει πως θέλει να τοποθετηθεί μέχρι τώρα. Η κυρία Μπίλτ. Μάλιστα, εφόσον οι σκιώδει εισηγητέ δεν επιθυμούν το λόγο, τότε φυσικά μπορούν και τα υπόλοιπα μέλη τη Επιτροπή να μιλήσουν. Η κυρία Σόιντροβα έχει το λόγο. Σα ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα και εγώ να ζητήσω χρόνο ομιλία. Ε, ναι, εφόσον δεν υπάρχει κάποιο σκιώδη. Σα ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πολύ τον εισηγητή για την έκθεσή του, η οποία είναι πολύ ικανοποιητική, ταυτόχρονα όμως και ασκή κριτική. Ο πολιτισμός είναι πάρα πολύ σημαντικός, γι' αυτό χαίρομαι πάρα πολύ με ε, το ότι υπογραμμίζεται ο κοινωνικός ε, και πολιτικός της ρόλος. Οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πάρα πολύ ε, σημαντικοί σημαντικό στοιχείο του πολιτισμού και είναι πολύ σημαντικό να είναι ευχαριστημένοι και ικανοποιημένοι με ε, τη στήριξη που δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση στον πολιτισμό. Σίγουρα μπορούμε να βελτιώσουμε πάρα πολλά τις ε, μεμονωμένες ε, πλατφόρμες, να στηρίξουμε τα σημεία επαφής. Αυτό φυσικά δεν είναι κάποια καινούργια ιδέα, όμως αξίζει τη στήριξή μας και οφείλουμε να το αναγνωρίσουμε ως κάτι πολύ θετικό. Επιπλέον, δύο σημαντικά σημεία. Η δημιουργική Ευρώπη, το Creative Europe, πρέπει να στηριχθεί ακόμα περισσότερο. Πολλοί μας έχουν ασκήσει κριτική στη διαδικασία. Λένε πως είναι περίπλοκη, χρονοβόρα. Γι' αυτό λοιπόν οφείλουμε να δούμε την κατάσταση και να την βελτιώσουμε. Ακριβώς επειδή δεν υπάρχουν αρκετά κονδύλια, θα πρέπει επίσης ε, να διατίθενται με όσο το δυνατόν περισσότερη διαφάνεια. Αυτό ήθελα να το τονίσω. Και επίσης, οφείλουμε να αναγνωρίσουμε ότι στην Ευρώπη υπάρχουν πάρα πολλές δραστηριότητες στα πλαίσια των, ε, της πολιτισμικής πρωτεύουσας ε, της Ευρώπης. Ε, για παράδειγμα το βραβείο Λούξ και διάφορες άλλες. Και αυτές τις εκδηλώσεις θα πρέπει να τις χρησιμοποιήσουμε συστηματικά για να προωθήσουμε την αξία του πολιτισμού. αυτές τις δράσεις μπορούν να τις αναλάβουν και να τις συντονίσουν και μεμονωμένα πόλεις και διάφορε, διάφοροι οργανισμοί, αλλά νομίζω πως καλύτερα θα ήταν να συνδυαστούν όλα αυτά έτσι ώστε μέσω της συνεργασίας να προωθήσουμε ε, όσο το δυνατόν περισσότερο τον πολιτισμό. Επίσης, η πολιτισμική, στα πλαίσια της πολιτισμικής κληρονομιάς θα μπορούσε να δημιουργηθεί ένα δίκτυο ε, το οποίο θα ε, χρηματοδοτηθεί Και επίσης, νομίζω πως ε, σε τελική ανάλυση θα πρέπει να δούμε ποια προγράμματα ε, λειτουργούν σωστά και ε, αυτά να τα στηρίξουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Κώστα έχει το λόγο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Γραμματικάκη για την εξαιρετική αυτή έκθεση που αποτελεί μια πολύ καλή βάση. Γιατί εμείς ως Επιτροπή θέλαμε να αντιδράσουμε στο κείμενο της Κομισιόν, γνωρίζοντας ότι η σημερινή ατζέντα που ξεκίνησε ε, την σημερινή εποχή ξεκινά το 2007. Έτσι λοιπόν με μία απόσταση 11 ετών θέτουμε σε νέα κίνηση μιας πιο ολιστικής και πλήρους στρατηγικής. Αυτό μας φαίνεται ένα σημαντικό βήμα προς τα μπρος. Και εκτιμώ πάρα πολύ τις προτάσεις και τις παρενέσεις του κυρίου Γραμματικάκη. Δεύτερο σχόλιο αυτή η ατζέντα και το αναγνωρίζει και η Κομισιόν συμπεριλαμβάνει πολλά από τα αιτήματα που συμπεριλαμβανόντουσαν και στις δικές μας εκθέσεις εφαρμογής των προγραμμάτων και ε, είχαμε ουσιαστικά ακολουθήσει τρεις-τέσσερις γραμμές. Η ε, πολιτιστική διπλωματία που έχει γίνει τώρα διεθνής διάσταση, η στρατηγική για την καιροτομία, για τους δημιουργικούς τομείς είναι στρατηγική για την ανάπτυξη το θέμα των πολιτιστικών αρμοδιοτήτων και καλλιτεχνικών ε, αρμοδιοτήτων ε, στο πλαίσιο της ψηφιακής στρατηγικής. Εδώ θα ήθελα να εμβαθύνουμε και για το ευρωπαϊκό έτος ε, της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς. Έχουμε λοιπόν τώρα με την ατζέντα μία δυνατότητα να έχουμε μία μακροπρόθεσμη στρατηγική η οποία ουσιαστικά καθιστά πιο εμφανές το γεγονό ότι μας λείπουν τα κονδύλια. Με τη Δημιουργική Ευρώπη βρισκόμαστε νομίζω στο 0,5% του ΑΕΠ. Εμείς έχουμε ζητήσει διοπλασιασμό και θα το ζητήσω και εγώ. Πρέπει να ζητήσουμε ακόμη περισσότερα κονδύλια, όπως είπε και ο συνάδελφο Μόργανο. Ίσως θα πρέπει να ζητήσουμε και περισσότερα κονδύλια και συνεργασία στο Horizon μεταξύ έρευνα και πολιτισμού και με την ψηφιοποίηση που σωστά θέτει ο κύριος Γραμματικάκη ως στόχο. Συμφωνώ 100% για την πύλη. Επίσης, είχαμε ζητήσει στο παρελθόν μία πύλη δική από την πλευρά της Κομισιόν, έτσι ώστε οι πολίτες να μπορούν να γνωρίζουν όλες τις ευκαιρίες. Εμείς δεν το έχουμε ακόμα σήμερα, αλλά νέου θέτουμε αυτό το αίτημα, αλλά και οι άνθρωποι αυτοί που μπορούν να συμμετέχουν σε αυτά τα προγράμματα κινητικότητα, είτε ε, προέρχονται από τρίτε χώρε είτε από ευρωπαϊκέ χώρε, να μπορούν να λαμβάνουν και μια κατάλληλη απάντηση. Να προσθέσω κάτι και κλείνω. Εκτιμώ ότι στην έκθεση γνωμοδότηση του κυρίου Γραμματικάκη ε, πρέπει να γίνει μια ε, πολύ συγκεκριμένη αναφορά, μια αναφορά στην μη καταλληλότητα των στατιστικών στοιχείων, ποιοτικών στατιστικών στοιχείων και της εγγενούς αξίας ε, των ποσοτικών στοιχείων. Ε, δηλαδή αυτό δεν ε, βοηθά τις χώρες να συγκριθούν, ούτε βοηθά την Κομισιόν να αναπτύξει μια λογική για να ενισχύσει τον θετικό αντίκτυπο. Ο αντίκτυπος είναι όχι μόνο τεχνολογικός, οικονομικός ή ψηφιακός. Η αντίκτυπος στην καινοτομία, αλλά αντίκτυπος κοινωνικής συνοχή και συμμετοχή σαν το 36% των πολιτών ποτέ δεν είχαν πρόσβαση στον πολιτισμό. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να το επιλύσουμε. Έτσι λοιπόν ζητάω από τον Γιώργο μήπως ρητά να προσθέσει μια ξεχωριστή διάσταση, μια αυτόνομη διάσταση για την καλλιτεχνική πολιτιστική αξία ε, και την ε, αναγνώριση της ιδιαιτερότητας ε, του πολιτιστικού τομέα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Uh, um, Ευχαριστώ και εγώ θα ήθελα να συγχαρώ τον εισηγητή για αυτήν την εξαιρετική έκθεση που καλύπτει ένα μεγάλο εύρος θεμάτων. Το θέμα της διαφορετικότητας της πολυμορφίας, η ευρωπαϊκή, ε, ο ευρωπαϊκός πολιτισμός και πριν ξεκινήσει, αν θέλετε, η μαζική μετανάστευση ουσιαστικά έχει αυτή τη διάσταση της πολυμορφίας και μιλάμε εδώ για πολιτισμό. Υπάρχει όμως και μια άλλη διάσταση που δεν είναι τόσο θετική η πολυμορφία και η διαφορετικότητα όσον αφορά και το θέμα της, του κοινωνικού, αν θέλετε, πολιτισμού. Χρειαζόμαστε κάποιες κοινέ ε, πολιτιστικές αξίες που να υιοθετούνται και να είναι κοινέ σε όλους η ελεύθερη έκφραση, η ισότητα των φύλων, η ισότητα και κάποιες αρχές οι οποίες ουσιαστικά θα πρέπει να γίνουν κοινέ κοινό αγαθό για όλους. Βλέπετε ότι σήμερα υπάρχουν στην Ευρώπη πληθυσμοί οι οποίοι προϋπήρχαν των μεταναστών και οι οποίοι διαμαρτύρονται, διαμαρτύρονται διότι θεωρούν ότι η συμπεριφορά και ο τρόπος ε, αντιμετώπισης αυτών που εισέρχονται στην Ευρώπη είναι διαφορετικός. Αυτή λοιπόν η διαμαρτυρία θα σταματήσει και θα ησυχάσουμε στην Ευρώπη αν υπάρξουν κοινά αγαθά και κοινέ αξίες. Uh, thank Η κυρία Σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ πραγματικά εκτιμώ την εργασία του συναδέλφου, του κυρίου Γραμματικά. Ε, πραγματικά έχει ενσωματώσει στην έκθεσή του και πολύ σημαντικές ε, ιδέες όπως την ελευθερία έκφρασης. Είναι εξαιρετικά σημαντικό αυτό. Η ελευθερία έκφρασης, η ελευθερία δημιουργίας ε, στον πολιτισμό, όλα αυτά τα οποία θα πρέπει να εκφράζονται με σαφήνεια και να προστατεύονται. Σήμερα το πρωί εδώ στο Κοινοβούλιο διοργανώσα μία συνάντηση με θέμα τις απειλές ε, προς τους δημιουργούς, προς τους καλλιτέχνες και τον καλλιτεχνικό κόσμο. Είναι εξαιρετικά σημαντικό λοιπόν το θέμα αυτό και για αυτούς οι οποίοι σήμερα ε, είναι πολιτική στην Ευρώπη, αλλά και για όλους αυτούς οι οποίοι νοιάζονται για τον πολιτισμό και τους καλλιτέχνες. Είναι πολύ σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε ότι σήμερα υπάρχουν πολύ σημαντικές ιδέες που ενσωματώθηκαν στην έκθεση αυτή. Σήμερα μιλάμε για πολιτισμό, μιλάμε όμως για δημιουργία και σε άλλους τομείς όπως τα μαθηματικά, η δημιουργικότητα, η περιέργεια, η επιστημονική διερεύνηση, οι αρχιτέκτονες παραδείγματο χάρη είναι κάτι μεταξύ του καλλιτεχνικού κόσμου και των μαθηματικών και της επιστήμης. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να δούμε ότι δεν υπάρχουν στεγανά, ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να αναφέρουμε να αναφερόμαστε στον πολιτισμό χωρίς να συμπεριλαμβάνουμε όλους αυτούς τους κόσμους της δημιουργικότητας. Σήμερα το απόγευμα λοιπόν Συζητούμε για τη σημασία των καλλιτεχνών, για την ε, δυνατότητα που πρέπει να τους παρέχουμε να ζουν από την ε, δημιουργία τους. Την επόμενη εβδομάδα θα ψηφίσουμε για τα πνευματικά δικαιώματα και θα πρέπει να στηρίξουμε τους καλλιτέχνες, να στηρίξουμε τους δημιουργούς οι οποίοι επαναλαμβάνω θα πρέπει να μπορούν να ζήσουν από τη δουλειά τους. Και σε καμία περίπτωση δεν θέλω να δεχτούμε μία αμερικανική κουλτούρα, έναν πολιτισμό ο οποίος θα προέρχεται από τις Ηνωμένε Πολιτείες. Ας στηρίξουμε λοιπόν το ευρωπαϊκό μας σχέδιο για τον πολιτισμό. Όπως ξέρετε, ο πολιτισμός έπαιξε πρωταρχικό ρόλο στην δημιουργία και την ολοκλήρωση της Ευρώπης και θα πρέπει να στηρίξουμε όλες τις πρωτοβουλίες, όλες τις προσπάθειες από τα πρώτα φεστιβάλ μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο το 1947, όταν ξεκίνησαν τα πρώτα φεστιβάλ. Πιστεύουμε στον πολιτισμό στην Ευρώπη, πιστεύουμε στην ειρήνη, πιστεύουμε στον διάλογο με τους γειτονές μας και όχι στην αντιπαράθεση. Γι' αυτό και το θέμα της στρατηγικής και της πολιτικής διπλωματίας είναι εξαιρετικά σημαντικό. Ας μην ξεχνάμε λοιπόν τι είναι η Ευρώπη και τι είναι το ευρωπαϊκό κοινό μας σχέδιο. Όλα αυτά πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι δεν είναι τυποποιημένα, ότι δεν είναι σταθερές αξίες οι οποίες δεν αλλάζουν, δεν μεταλλάσσονται. Είναι σημαντικό να συμπεριλάβουμε τα νέα πραγματικότητα, την πολυμορφία, την πολυγνωσία, το ότι η Ευρώπη σήμερα ενσωματώνει και άλλους πολιτισμούς, ενσωματώνει και το Ισλάμ, και μην ξεχνάμε ότι η Αλάμπρα στην Ισπανία είναι ένα πανέμορφο οικοδόμημα το οποίο δημιουργήθηκε από τους Άραβες και ενσωματώθηκε στον ευρωπαϊκό πολιτισμό. Το Ισλάμ λοιπόν δεν είναι κάτι καινούριο στην Ευρώπη. Εδώ και χιλιάδες χρόνια γνωρίζουμε το Ισλάμ και κάποιοι θα πρέπει να το ξεπεράσουν. Thank you. The next is... Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στον κύριο Γραμματικάκη, διότι όπως άκουσα και στην ακρόαση τον Ιούλιο, αυτή η νέα ατζέντα θα πρέπει να αποτελεί δανεική ευκαιρία διότι αυτό που ενώνει τους πάντες στην Ευρώπη στην ουσία είναι ο πολιτισμός. Θα πρέπει λοιπόν να δημιουργηθεί μία νέα πλατφόρμα που θα περιέχει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες. Αυτό είναι κέρια σημασία, διότι σε τελική ανάλυση πρέπει αυτήν τη νέα ατζέντα να τη δούμε και στο πλαίσιο της τεχνολογίας, να δούμε ποιες δυνατότητες τεχνολογικά έχουμε. Τώρα, σε ό,τι αφορά αυτά που υπόθηκαν, θα ήθελα και εγώ να δώσουμε έμφαση στην ελευθερία έκφρασης, γιατί αυτό είναι στο κέντρο ε, του οτιδήποτε σημαίνει ο πολιτισμός. Ο πολιτισμός δεν μπορεί να θεωρηθεί πολιτισμός χωρίς την ελευθερία της έκφρασης. Και εγώ στη δική μου χώρα όταν βλέπω οποιαδήποτε παρέμβαση στον πολιτισμό, είτε αυτό είναι επιλογή καλλιτεχνών για συγκεκριμένες εκδηλώσεις είτε κάτι άλλο, παρατηρώ ότι τέτοιες παρεμβατικές ενέργειες πλήττουν σφοδρά τον πολιτισμό. Μετά, να δούμε για την κινητικότητα, διότι ε, ένας καλλιτέχνης όταν προέρχεται από μια μικρή χώρα όπως η Μάλτα πρέπει να έχει περισσότερες ευκαιρίες να ταξιδέψει και να δείξει τη δουλειά του, να παρουσιάσει το έργο του. Το κενό αξιών επίσης είναι κάτι που πρέπει να εξετάσουμε. Πρέπει να δούμε τι γίνεται με τα, δικαιώμα, με τα πνευματικά δικαιώματα, και να σας πω ότι έχω συναντηθεί με διάφορους ε, φορείς και εκεί οι καλλιτέχνες μου εξέφρασαν ε, τα παράπονά τους για την αποζημίωσή τους. Πολλές φορές ε, δεν αποζημιώνονται ούτε καν για τα έξοδα τα οποία πληρώνουν οι ίδιοι. Δεν ανταμείβονται για τον κόπο τους, για τη δημιουργικότητά τους. Σίγουρα λοιπόν αυτή είναι μια πτυχή που δεν πρέπει να παραγνωρίζουμε. Επίσης υπάρχει και μια άλλη σημαντική διάσταση Σίγουρα η ευρωπαϊκή διάσταση είναι κάτι που πρέπει να προωθούμε και να μας κάνει υπερήφανους, διότι διαφορετικά θα γίνουμε όλοι οι Αμερικάνοι. Αυτό πάει κυρίως στον χώρο του κινηματογράφου. Θα ήθελα να βλέπουμε περισσότερες ευρωπαϊκές ταινίες, να προβάλλονται σε σχολεία, να δίνουμε περισσότερο χώρο στο ευρωπαϊκό σινεμά. Ε, εδώ θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε και την ε, οδηγία για τα οπτικοακουστικά μέσα, όμως δεν πρέπει να στεκόμαστε μόνο σε αυτή. Πρέπει η πολιτική να είναι ευρύτερη. Ε, δεν ε, είναι ο κινηματογράφος μόνο το Hollywood ή το Bollywood, είναι και η Ευρώπη. Και πρέπει να δούμε λοιπόν τι γίνεται εντός της περιοχής μας. Επίσης, θα ήθελα να πω ότι για τους Ευρωπαίους ταυτότητα και η πολιτισμική πολυμορφία είναι πάρα πολύ σημαντική και είναι εργαλείο για το διαπολιτισμικό διάλογο. Τέλος, γίνεται λόγος για καινοτομία, οπότε ας επενδύσουμε και στους καινοτόμους, στην οποία περίπτωση καινοτόμοι είναι καλλιτέχνες. Πρέπει να δείξουμε την ε, εκτίμησή μας στους καλλιτέχνες και το έργο τους, γι' αυτό και οφείλουμε να εξασφαλίσουμε μία αξιοπρεπή διαβίωση και αναγνώριση του έργου τους. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Πρόεδρε, σημειώνω αυτό που λέτε ότι δεν παίρνουμε αρκετά το λόγο. Υπάρχει μεγάλη απουσία μελών εδώ στην Επιτροπή. Εγώ κάθε φορά παίρνω το λόγο, σήμερα όμως δεν είμαι πολύ καλά. Πιστεύω μάλιστα ότι θα αναγκαστώ να φύγω από την αίθουσα. Βεβαίως, ε, εάν θεωρείτε ότι πρέπει οπωσδήποτε να πάρω το λόγο και να εκφράσω την απόψή μου, θα το κάνω, αλλά ε, πραγματικά δεν νιώθω καλά. Θέλετε οπωσδήποτε να εκφράσω την άποψή μου. Έχετε δικαίωμα να πάρετε το λόγο ή να σιωπήσετε. Εγώ καλώ όλους τους εκπροσώπους ε, των ομάδων και τώρα θα δώσω το λόγο και στην Επιτροπή. Θέλετε να πάρετε το λόγο. Thank you. Good afternoon. Um, I too would like to uh, thank. Um, και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή, τον κύριο Γραμματικάτη, για την έκθεσή του. Είναι εξαιρετικά πλήρης και πραγματικά συμβαδίζει με τις προτάσεις ε, της ε, Επιτροπής που υιοθετήθηκαν το Μάιο. Γίνονται κάποιες εκκλήσεις προς την Επιτροπή, θα συμφωνήσουμε στις περισσότερες. Εξάλλου οι απαντήσεις βρίσκονται και στο ίδιο το έγγραφο. Μιλάμε και για το μέλλον του προγράμματος. Υπάρχουν αντικείμενα που σίγουρα θα αποτελέσουν ε, σημεία διαπραγμάτευσης ε, για άλλα θέματα όπως το Creative Euro παραδείγματος χάρη. Καταλαβαίνω τις ε, προτάσεις κάποιων μελών του Κοινοβουλίου όσον αφορά ένα συγκεκριμένο τόπο όπως μια συγκεκριμένη θηρίδα, ένα one-stop shop για την παροχή περισσότερων πληροφοριών με πιο συγκεντρωτικό τρόπο. Το θέμα τώρα της χρηματοδότησης όλων αυτών των προγραμμάτων, όπως της πολιτιστικής κληρονομιάς, υπάρχουν επίσης και οι αρμόδιοι για τα προγράμματα αυτά, οι οποίοι ήδη λειτουργούν και εργάζονται στις χώρες μέλη. Προσπαθήσαμε επίσης να ενσωματώσουμε πολιτιστικά προγράμματα και σε πολλούς άλλους τομείς όπου δραστηριοποιείται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Να ενσωματώσουμε δηλαδή συνιστώσεις πολιτιστικές και σε άλλα προγράμματα. Βεβαίως μπορούμε να κάνουμε πολύ παραπάνω και με μεγάλη χαρά θα εξετάσουμε τις προτάσεις για να βελτιώσουμε τη δράση μας στο μέλλον. Αυτή η προσπάθεια αυτής της νέας ε, τέντας για τον πολιτισμό κάνει και ένα είδος απολογισμού όλων των προγραμμάτων, ένα κατάλογο όλων των προγραμμάτων και βεβαίως υπάρχει και το τρισέλιδο έγγραφο το οποίο περιέχει ένα μεγάλο αριθμό πληροφοριών και στοιχείων για όλα αυτά τα προγράμματα το οποίο ακολουθεί την πρότασή μας. Όσον αφορά την πολυμορφία των ε, μέσων και το βαθμολόγιο το οποίο ζητήσατε, νομίζω ότι υπάρχει ένας τρόπος σύγκρισης ε, και παρακολούθησης της πολυμορφίας στα μέσα. Νομίζω ότι αυτό μπορείτε να το βρείτε εξάλλου και στο πρόγραμμά μας, το οποίο μπορείτε να κοιτάξετε το θέμα της πολιτιστικής πολυμορφίας, κάτι που πραγματικά μας απασχολεί εδώ και πολλά χρόνια στην Επιτροπή και έχουμε θέσει και πολύ συγκεκριμένους μεθοδολογικούς στόχους. Σας ευχαριστώ πολύ. Thank you too. Σας ευχαριστώ. Να δώσω το λόγο στον εισηγητή για τρία λεπτά για τις τελικές του παρατηρήσεις. Είμαι πολύ σύντομος. Ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους για τις πολύ χρήσιμες παρατηρήσεις τους. Ειλικρινά το πιστεύω. Για την κυρία Στόλονταβα ήθελα να πω ότι η δημιουργική Ευρώπη πράγματι υποφέρει και ως προς τις διαδικασίες και τονίζω στην έκθεση ότι πρέπει να γίνουν απλούστερες εκτός από τη χρηματοδότηση. Για την κυρία Κώστα είναι πολύ θετικό ότι αυτή η έκθεσή μου περιλαμβάνει όπως είπε πολλά από τα αιτήματα της Επιτροπής Πολιτισμού, της δίνει μεγαλύτερο κύρος. Είναι επίσης εμφανές ότι λείπουν τα κονδύλια παντού και η αναφορά στα στατιστικά στοιχεία συμφωνώ ότι πρέπει να έχει και ποιοτικέ παραμέτρους. Ο κύριος Φλίν μίλησε πολύ εύστοχα για τις κοινέ πολιτιστικές αξίες Αυτές νομίζω περιλαμβάνουν και τις αξίες των προσφύγων ή των μεταναστών οι οποίοι ενσωματώνται στην ευρωπαϊκή κουλτούρα και η κυρία Ward τόνισε την ελευθερία της έκφρασης όπως το τονίζουμε και εμείς στην έκθεση ε, και για πρώτη φορά επεσήμανε τον κίνδυνο θα έλεγα εγώ από μια επελάβνουσα, από μια δυναμική ευρωπαϊκή, αμερικάνικη κουλτούρα το τόνισε και ο κύριος Ζάμιτ αυτό και ο κύριος Ζάμιτ επίσης τόνισε όπως η έκθεσή μου την έφαση στην αξία του πολιτισμού και επίσης τα πνευματικά δικαιώματα που αποτελούν ένα κυρίαρχο μέλος της ε, εκθέσεώς μου. Ευχαριστώ επίσης τον εκπρόσωπο της Κομισιόν γιατί έδειξε από την αρχή το συνεργατικό του πνεύμα και επεσήμανε σημεία που και εμείς έχουμε επισημάνει στην έκθεση και θα ήθελα να καταλήξω, κυρία Πρόεδρε, με μια ιδέα που είχα, δεν την έβαλα ακόμα στην έκθεση, ε, γιατί ήθελα να δω τις αντιδράσεις των συναδέλφων. Η ιδέα που έχω και παρακαλώ να τη σκεφτείτε και να να το κάνουμε σαν τροπολογία είναι όχι μόνο να υπάρχει έτος πολιτιστικής κληρονομιάς, αλλά θα το πω πολύ γενικά να υπάρχει και έτος πολιτιστικής προσωπικότητας. Δηλαδή ενός ανθρώπου που θα συνδυάζει με το έργο και την απίσυσή του τις ευρωπαϊκές αξίες. Να σας πω μόνο μερικά ονόματα που εγώ θα βράβευα μέσα σε αυτό το σημείο για να τα σκεφτείτε. Λεωνάρδο Νταβίντσι, ο Όμηρος ή ο Πλάτων βέβαια, ο Σέξπιρ, ο Γκέτε, ο Πικάσο, ο Μπετόβεν ή ο Μόζερτ, ο Βίσεντ Βακόγκ, ο Μιτσελάγγελο. Η ο πλατων βεβαια ο σεξπιρ ο γκετε ο πικασο ο μπετοβεν η ο Μόζελ, ο βισεντ βακογκ ο μιτσελαγγελο η ιδεα μου λοιπόν είναι να αποκτήσουμε ακριβώς για την προβολή του πολιτισμού και το θεσμό της πολιτιστικής προσωπικότητας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κυρία Γραμματικάκη για αυτή την πολύ καλή ιδέα και για τα σχόλιά σας. Νομίζω ότι είναι εξαιρετική ιδέα. Η Ουγγαρία έχει ένα είδος συστήματος, φάση του οποίου αφιερώνουμε ένα χρόνο σε μια διάσημη προσωπικότητα, σε έναν μεγαλοποιητή ή καλλιτέχνη, παραδείγματο χάρη στη χώρα μας. Και διοργανώνουμε διάφορες εκδηλώσεις σε σχολεία ή προσπαθούμε να δημοσιεύσουμε τα έργα τους. Λοιπόν, να σας υπενθυμίσω ότι η προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών είναι στις 12 Σεπτεμβρίου το μεσημέρι, 12 το μεσημέρι και θα ψηφίσουμε στις 20 Νοεμβρίου στην Επιτροπή μας. Ολοκληρώνουμε λοιπόν αυτό το σημείο και περνάμε στο επόμενο που είναι η εξέταση του σχεδίου γνωμοδότησης που αφορά την ενδιάμεση έκθεση για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-2027. Η κυρία Κάμερβερτ είναι η συγγήτρια. Προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών είναι η 6η Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα. Η ψηφοφορία στην Επιτροπή μας 10 Οκτωβρίου και στην Αρμόδια Επιτροπή η budget θα ψηφίσει στις 5 Νοεμβρίου. Τα επόμενα τέσσερα τιμία στην ημερήσια διάταξή μα όλα σχετίζονται με σχέδια γνωμοδοτήσεων που αντιδρούν στην ε, πρόταση της Κομισιόν για το επόμενο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο και τις αντίστοιχε νομοθετικές προτάσεις για συγκεκριμένα προγράμματα. Το πρώτο σχέδιο γνωμοδότησης που θα συζητήσουμε αφορά το ίδιο το πολιτες δημοσιονομικό πλαίσιο. Ο κανονισμός PDPE έχει στηθεί υπό, υιοθετείται μάλλον υπό τη διαδικασία συνένεσης δυνάμει του άρθρου 312 της συνθήκης δηλαδή το Κοινοβούλιο μπορεί να εγκρίνει ή να απορρίψει τον προτινόμενο κανονισμό. Η γνωμοδότηση σχετίζεται με την ενδιάμεση έκθεση και αποτελεί απάντηση στην πρόταση για το πολιτές του Πλαίσιο της Δευτέρας Μαΐου 2018. Σκοπεύει να παρουσιάσει τη θέση του Κοινοβουλίου για τις κύριες δημοσιονομικές πτυχές ε, των αριθμών του πολιτές δημοσιονομικού πλαισίου. Λείπει δυστυχώς η συγγήτρια σήμερα, επομένως η κυρία Τζούλι Γουόρντ θα την εκπροσωπήσει. Θα ήθελα να της δώσω το λόγο. Λοιπόν, ε, θα διαβάσω εδώ τι λέει η Πέτρα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους ε, τους σκιώδες, τη γραμματεία της Επιτροπής, ε, τους συμβούλους και τους βοηθούς για την πολύ εστιασμένη δουλειά που έχουμε κάνει μέχρι σήμερα και μπορούμε να πούμε και για όλους τους φακέλους που έχουν να κάνουν με το πολιτισμό-συνομικό πλαίσιο. Πιστεύω ότι είναι η ορθή ευκαιρία να τονίσουμε εκ νέου ότι εμείς ως Επιτροπή Πολιτισμού περιμένουμε περισσότερες προσπάθειες ό,τι αφορά το Εράσμος και τη Δημιουργική Ευρώπη υπό το τομέα που καλείται επενδύοντα στους ανθρώπου, Επαναλαμβάνω, τα αιτήματά μα να τριπλασιαστούν τα κονδύλια τουλάχιστον για το Erasmus και να διπλασιαστούν τουλάχιστον τα κονδύλια για το Creative Europe και να αυξηθούν τα κονδύλια για τα μέτρα ηθαγένεια και το Ταμείο Αξιών. Επιμένω, όλες οι πολιτικές αποφάσεις ε, θα πρέπει να βασίζονται στη νομική βάση ή να χρησιμοποιούνται τα εξουσιοδότηση πράξη, αλλά να μην ε, διευρύνεται το πεδίο εφαρμογή των εκτελεστικών πράξεων όταν ε, περιέχονται πολιτικέ επιλογέ. Καθώ το σχέδιο τη έκθεση έχει περιορισμένο χώρο, συζητήσαμε με τη Γραμματεία και του Σκιώδη Ηγητή κάποιε πιθανέ κοινέ τροπολογίε. Οι Σκιώδη και οι Σύμβουλοι Πολιτική ε, ε, ενημερώθηκαν για την τελευταία κατάσταση την ε, προηγούμενη Παρασκευή και ε, καλείστε να σχολιάσετε επί αυτών των κοινών τροπολογιών. Αυτό να το κάνετε μέχρι την Τρίτη το μεσημέρι παρακαλώ. Με τις κοινέ τροπολογίες προτείνω την ενδυνάμωση του σημείου ήθελα να τονίσω με σαφήνεια τι περιμένουμε ως προς τις συνέργειες μεταξύ διαφορών προγραμμάτων. Ακόμη και με το νομικό κείμενο δεν είναι σαφές ε, πόσο η συνέργεια θα υλοποιηθεί και θα διατηρηθεί στην πράξη. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε την αναγκαιότητα μια ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία ε, που τα δημόσια κονδύλια θα πρέπει να υπηρετούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο την, ε, με την επόμενη πράσινη εβδομάδα στο Στρασβούργο για την αποστολή στο Σαν Φρανσίσκο, Αν τα λάβουμε όλα αυτά υπόψη. Θα ήθελα να έχουμε μικρή προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών. Ε, η λήξη είναι 6 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα. Όμως ε, έτσι θα μπορέσουμε να ψηφίσουμε στις 10 Οκτωβρίου, αν έχουμε περισσότερο χρόνο για να βρούμε συμβιβαστικές τροπολογίες βάσει αυτού του διαγράμματος. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Ward. Και κάτι πολύ σημαντικό. Στις 11 Ιουλίου οι συντονιστές αποφάσισαν τα ακόλουθα. Οι τροπολογίες θα κατατεθούν μόνο στην αγγλική γλώσσα. Θα ήθελα λοιπόν να σας παρακαλέσω όλους να το σημειώσετε. Και τώρα θα δώσω το λόγο στους κοιόδης εισηγητές και στον κύριο Στρογεύσκη πρώτα. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ξεκινήσω με ένα σχόλιο ε, πάνω στην ε, προηγούμενη ψηφοφορία για το 2019. Νομίζω πως ε, παρότι πήγαν όλα καλά, δεν ήταν εύκολο να ε, συμβιβαστούμε στις τροπολογίες. Νομίζω το είδαμε αυτό. Βλέπουμε ποιες τροπολογίες ε, ψηφίστηκαν από μεγάλη πλειοψηφία. Ήταν εκείνες οι οποίες κατατέθηκαν από τις μεγαλύτερες πολιτικές ομάδες. Οι δικές μου, οι τροπολογίες κυρία Τρούπελ και του κυρίου Μπάμπατς έχουν εγκριθεί Και αυτές οι τροπολογίες κάλυπταν όλα τα επίμαχα σημεία στην έκθεση. Τώρα βέβαια ελπίζω αυτή η συνένεση να μεταφερθεί και στην συζήτηση για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Να πω ότι επί της αρχής δεν διαφέρουμε στις απόψεις. Μόνο στην περίπτωση του εράσμους πλάση υπάρχουν κάποιες ε, διαφορές. Στο τέλος της, ε, περίοδου, της προγραμματικής περίοδου θα έπρεπε η χρηματοδότηση να τριπλασιαστεί. Γι' αυτό θα σας παρακαλέσω όλους να, ακολουθήσετε, να με ακολουθήσετε σε αυτή την άποψη. Έπειτα, το πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη υποχρηματοδοτείται συστηματικά και υπάρχουν πάρα πολλές καλές προτάσεις οι οποίες δεν μπορούν να υλοποιηθούν ακριβώς επειδή δεν υπάρχει χρηματοδότηση. Χρειάζεται λοιπόν διεύρυνση και του προγράμματος Δημιουργική Ευρώπη. Για την ακρίβεια ζητούμε διπλασιασμό της χρηματοδότησης. Και να τονίσω ότι ακόμα και ο διπλασιασμός της χρηματοδότησης δεν θα είναι αρκετός για να χρηματοδοτήσει όλα τα αξιόλογα project. Οι αιτήσει λοιπόν που εγκρίνονται και αυτές που στην ουσία πραγματικά υλοποιούνται απέχουν πολύ μεταξύ τους. Τώρα, Έχουμε συζητήσει το θέμα αυτό με πολλές αφορμές. Η κυρία Κώστα, η κυρία Κάμερ Εύερτ και η κυρία Φερχάιεν, ο κύριος Μόργαν, όλοι οι συνάδελφοι είπαν λίγο πολύ ότι τα πάντα χρειάζονται βελτίωση. Δηλαδή, τι εννοώ, πρόθεση, επικοινωνία, ενημέρωση, και οτιδήποτε συνδέεται με την ψηφιακή διάσταση αυτών. Τέλος, είναι πολύ σημαντική η ευελιξία στην χρηματοδότηση και στην διάθεση κονδυλίων. Υπάρχουν δικαιούχοι οι οποίοι περιμένουν τη χρηματοδότηση, η χρηματοδότηση που λαμβάνουν είναι πολύ μικρή, είναι τα οικονομικά τους πολύ σφιχτά και στο τέλος έχουν να αντιμετωπίσουν και τεράστια γραφειοκρατία. Πρέπει λοιπόν να προσέχουμε οι κανόνες να μην γίνουν τόσο αυστηροί που να μην μπορούν να προσαρμοστούν στις, ε, αλλά στις ε, ανάγκες της νέας γενιάς. Αυτά εν συντομία, δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο, γι' αυτό και ζητήσαμε τις τροπολογίες στα αγγλικά, όμως νομίζω πως πρέπει να αξιοποιήσουμε το χρόνο που έχουμε ως το δυνατόν περισσότερο για να καταλήξουμε σε μια καλή γνωμοδότηση. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εγώ. Η κυρία Τρούπελ έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ. Μόλις γύρισα από το Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας και συγγνώμη που άργησα, αλλά το αεροδρόμιο Βρυξέλλες ε, είναι χάλια, περίμενα μισή ώρα πάρω τη βαλίτσα μου. Και το Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας πραγματικά είναι μια διοργάνωση που νιώθει κανείς την καρδιά του ευρωπαϊκού ε, πολιτισμού. Η Βενετία είναι και μια πανέμορφη πόλη, υπάρχει λοιπόν ήδη το σκηνικό ε, Αυτόν που θα σας πω τώρα για τον πολιτισμό και για τη δημιουργική Ευρώπη και για το γιατί πρέπει να δώσουμε έμφαση σε αυτά. Θεωρώ λοιπόν ότι αν δει κανείς το τοπίο στην Ευρώπη θα παρατηρήσει ότι απειλείται ο πολιτισμός. Ο πολιτισμός που στηρίζει την πολυμορφία. Νομίζω πως κινδυνεύουμε να επιστρέψουμε στην έννοια της πόλης κράτους από την ε, ευρωπαϊκή ταυτότητα. Και μάλιστα ακούστηκε στην Ολομέλεια να, ότι εντάξει δεν χρειάζεται να ξεφορτωθούμε όλα αυτά τα πολιτισμικά διότι οι μόνοι που παράγουν πολιτισμό αυτή τη στιγμή είναι οι Γάλλοι. Όχι, όχι. Νομίζω πως ε, πρέπει να δούμε τη γενικότερη εικόνα. Ο πολιτισμός και η πολιτισμική ταυτότητα απειλείται και θεωρώ πως ε, εφόσον η δική μας Επιτροπή, η Επιτροπή μας Πολιτισμού έχει δείξει τη δυσαρέσκειά της με τόσο έντονο τρόπο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να δράσει. Θα πρέπει να δράσει όμως πώς, μειώνοντας τη χρηματοδότηση από άλλους τομείς, τη γεωργία για παράδειγμα, και εκεί θα γίνει η μεγάλη μάχη. Είναι μεγάλα τα συμφέροντα που παίζονται. Γι' αυτό, εάν θέλουμε να είμαστε ε, να επιτύχουμε, τότε θα πρέπει να προωθήσουμε την αξία του πολιτισμού ως ε, ένα μέσο χειραφέτησης ε, των νέων και των πολιτών εν γέννη. Ο πολιτισμός ε, είναι κάτι που φτάνει σε όλους τους πολίτες, φτάνει ιδιαίτερα στους νέους, γι' αυτό λοιπόν και πρέπει να του δώσουμε την απαραίτητη έμφαση. Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό και συνεισφέρει ιδιαίτερα σε αυτό. Γι' αυτό πρέπει να ε, το στηρίξουμε, καθώς και να στηρίξουμε το έργο που γίνεται στην επαρχία. Όπως είπατε και εσείς, διπλασιασμός του Creative Europe δεν είναι αρκετός, όμως θα δώσει ένα καλό μήνυμα. Ε, νομίζω, βέβαια πως δεν είναι διπλασιασμός, αλλά 30% αύξηση. Δεν ξέρω πώς το έχει φτιάξει εκεί ο Έτινγκερ. Αλλά εμείς ως Επιτροπή οφείλουμε να αναγνωρίσουμε το παιχνίδι αυτή τη στιγμή. Είναι παιχνίδι εξουσίας, πρέπει να αναλάβουμε τους ρόλους μας και να ε, προωθήσουμε το συμφέρον του πολιτισμού. Η διαπραγματευτική ομάδα νομίζω έχει δύσκολο έργο μπροστά τη με το Συμβούλιο. Οι διαπραγματεύσει θα είναι πολύ δύσκολε, ίσω οι δυσκολότερε των τελευταίων δεκαετιών, διότι υπάρχουν πολλέ κυβερνήσει που δεν είναι και τόσο ε, υπέρ της Ευρώπης και θα θέλουν να κρατήσουν τα χρήματα για ε, δικά τους έργα. Θα ήθελα λοιπόν να πω και εγώ στον κύριο Στρογεύσκη ότι ως Επιτροπή πρέπει να δείξουμε ε, πυγμή και σταθερότητα έτσι ώστε να μπορούμε να υπερασπιζόμαστε τα συμφέροντά μας και γι' αυτό είναι υπέρ όλων μας να βρεθεί συμβαστική λύση. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Κώστα έχει το λόγο. Θα ήθελα να αναφερθώ όσο είπε η συνάδελφος ε, Τρούπ ε, προηγουμένως ε, γιατί και εμείς εξ της Κομισιόν εξ της Επιτροπής μας δίνουμε μεγάλη σημασία στο φεστιβάλ της ε, Βενετίας. Νομίζω ότι υπάρχει πολύ μεγάλη ανάγκη για την Ευρώπη για να προχωρήσει το ευρωπαϊκό πρόγραμμα, να τροφοδοτείται από ελευθερία, καλλιτεχνική ελευθερία έκφρασης και από πολιτισμό. Τώρα, ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία θα πρέπει να αναρωτηθούμε. Όλοι είμαστε πεπισμένοι σε βάθος ε, ότι η Ευρώπη ε, αποτελεί μια αξία. Αυτή είναι τώρα, ε, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο αμφισβητείται, τίθεται υποσυζήτηση. Ε, τώρα, ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Ε, δεν θα έπρεπε να ε, μιλάμε μόνο γι' αυτό, αλλά κάθε project θα έπρεπε να έχει κάτι που να φέρνει αξία στην Ευρώπη και στο ευρωπαϊκό project. Εμείς ε, θα πρέπει να έχουμε κατά νου τι θα συμβεί στο επόμενο πολιτές δημοσιονομικό πρέσιο. Κρατώ τη βάση ε, της πρότασης της Πέτρα, αποτελεί μια καλή βάση και θέλω να απογραμμίσω τα εξή. Καταρχήν, Υπάρχει ένα μεγάλο ερώτημα που αφορά το ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ως συνομοθέτη. Πώς θα γίνει πιο ισχυρός ε, στην ε, μακροπρόθεσμη προοπτική, γιατί θα έχουμε και πολύ μεγάλες αλλαγές τα επόμενα 7 χρόνια. Συμφωνώ λοιπόν με την πρόταση που πρέπει να γίνει από την Επιτροπή μας, αλλά και από όλο το Κοινοβούλιο. Εμείς να προτείνουμε μία ρήτρα αναθεώρησης υποχρεωτική ενδιάμεση ρήτρα αναθεώρησης ε, που ουσιαστικά θα θέσει μια νέα εστίαση στις προοπτικές του πολιετές δημοσιονομικού πλαισίου. Γιατί εμείς μπορούμε να δεκτούμε τις ε, ε, εκτελεστικές πράξεις όταν μιλάμε για την ενεργοποίηση ενός κοινού προγράμματος. Αλλά αν μιλάμε για τη θέση νέων πολιτικών προτεραιοτήτων, τότε εμείς πρέπει να συμμετέχουμε. Αυτό είναι κεντρικό θέμα. Μας ε, αρέσει επίσης ότι η Κομισιόν, ε, τουλάχιστον η ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑ Πολιτισμού, προβλέπει πολύ περισσότερο κάποιες ε, συνέργειες μεταξύ των διάφορων προγραμμάτων με μεγαλύτερη δυνατότητα ενοποίησης των πόρων και των ευκαιριών. Βέβαια, στην πράξη κάτι τέτοιο είναι πάρα πολύ δύσκολο. Οι μηχανισμοί που προβλέπονται είναι πολύ light, ελαφρύ. Έτσι λοιπόν θα πρέπει να έχουμε διαφανείς και αποτελεσματικούς μηχανισμούς προς αυτή την κατεύθυνση. Τρίτον, πιστεύω ότι είναι προφανές τα αιτήματά μας, επί των οποίων πιστεύω η Επιτροπή Προϋπολογισμού ε, να τις λάβει υπόψη, μας το έχει υποσχεθεί ο εισηγητής, ελπίζουμε να συνάδει με τη γραμμή μας, όλες οι πολιτικές ομάδες θα πρέπει να το ζητήσουν από τους συναδέλφους της Επιτροπής εκείνης ε, προκειμένου ε, να διατηρήσουμε τη δέσμευσή μας απέναντι στους νέους για να έχουμε τριπλά κονδύλια για το Εράσμους και να μην έχουμε μόνο 0,5 των κονδυλίων για την ε, δημιουργική Ευρώπη. Σε μια τέτοια κρίση που διανύει η Ευρώπη αυτό είναι απολύτως ουσιώδες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Julie Βόρτ. Θα ήθελα να πω κάτι πιο προσωπικό. Να ευχαριστήσω καταρχήν την Πέτρα για το εξαιρετικό αυτό σχέδιο έκθεσης και γιατί πραγματικά είναι πάρα πολύ σημαντικό να δούμε το θέμα της παιδείας, της εκπαίδευσης των πολιτών, άτυπης αλλά και τυπικής. Είναι κάτι που φυσικά αντιμετωπίζουν τα κράτη-μέλη, είναι δική τους αρμοδιότητα, αλλά πρέπει να προετοιμάσουμε τους νέους πολίτες, τους νέους Ευρωπαίους, όσον αφορά πολλές δεξιότητες όπως η δυνατότητα σύγκρισης, κρίσης, ηγετικών ε, πρωτοβουλειών, δράσεις ε, σε συλλογικό και ατομικό επίπεδο. Και βεβαίως ξέρω ότι αυτό μπορούμε να το κάνουμε μέσω του πολιτισμού. Είναι πολύ σημαντικό αυτό και εγώ από την προηγούμενη δράση μου, πριν πω στην πολιτική, έχω την απόλυτη υπεποίθηση ότι μπορούμε να το κάνουμε αν δεν επενδύσουμε στους νέους, στον πολιτισμό, αν δεν ε, επενδύσουμε με κάθε τρόπο στην ε, χειραφέτηση των νέων μας, αν δεν διαθέσουμε πόρους, ενέργεια και χρόνο στην ε, καλλιέργεια των νέων μας, νομίζω ότι θα χάσουμε το στοίχημα του μέλλοντος. Ποιος θέλει να πάρει το λόγο για την Επιτροπή? Euh, Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σημειώνει όλα τα σχόλιά σας, ιδιαίτερα αυτά που αφορούν την ε, εκπαίδευση, τους νέους, τον πολιτισμό. Σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα για όλα αυτά που προτείνετε, το διπλασιασμό, τον τριπλασιασμό των προγραμμάτων Erasmus και Europe Creative και για τη στήριξή σας ε, για περισσότερη χρηματοδότηση στον προϋπολογισμό για προγράμματα πολιτιστικά. Όσον αφορά τα πολυετή χρηματοδοτικά σχέδια, βεβαίως και θέλουμε να αυξήσουμε την αποτελεσματικότητα της χρηματοδότησής μας, αλλά με μεγάλη ε, αυστηρότητα όσον αφορά την ε, προστιθέμενη αξία αυτών των επενδύσεων. Θέλουμε να είμαστε ρεαλιστές, να στηρίζουμε τις νέες προτεραιότητες, αλλά και προτεραιότητες υπάρχουσες, οι οποίες πραγματικά θα πρέπει να συνεχίσουμε να στηρίζουμε, παρόλη την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου. Η καινοτομία, η ψηφιακή οικονομία, ο πολιτισμός είναι τομείς εξαιρετικά σημαντική για τις νέες γενιές. Γι' αυτό και αποτελούν προτεραιότητες. Ευχαριστούμε πολύ, διότι όλοι αναφερθήκατε στην 30η επιτυχία του προγράμματος Εράσμους. Γι' αυτό και αποφασίσαμε να ενισχύσουμε την κινητικότητα των νέων και σε άλλους τομείς, όχι μόνο δηλαδή για τους φοιτητές, αλλά και για άσκηση, μαθητεία και άλλου είδους ανταλλαγές. Θέλουμε την ίδια ώρα να δίνουμε στοιχεία που να αναφέρονται σε πραγματικές τιμές, πραγματικούς αριθμούς δηλαδή, του 2018, για να βοηθήσουμε την συγκρισιμότητα των στοιχείων. Με αυτόν τον τρόπο νομίζω ότι είναι πιο κατανοητός ο προϋπολογισμός και ο ετήσιος ο οποίος όπως ξέρετε ψηφίζεται με αυτόν τον τρόπο την ίδια ώρα ξέρετε ότι υπάρχουν ε, δύο τρόποι παρουσίασης των τιμών καθώς και ο υπολογισμός, συνυπολογισμός ε, του πληθωρισμού η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να υπάρχει διαφάνεια στην παρουσίαση των ε, ποσών και των στοιχείων των αριθμητικών δίνουμε ακριβώς τις ε, τιμές, ε, σε σταθερές τιμές, σε τρέχουσες τιμές για την αύξηση δε των ποσών βλέπετε συν 122 και για το Creative Europe συν 34%. Παρουσιάζουμε επίσης τους διαφορετικούς τρόπους χρηματοδότησης. Προσπαθήσαμε να βελτιώσουμε τον τρόπο παρουσίασης των στοιχείων βάσει των νομοθετικών δυνατοτήτων που έχουμε χρησιμοποιώντας μεθόδους όπως το blending και διαφορετικές νομικές βάσεις για να αυξήσουμε την αποτελεσματικότητά μας. Η νέα αρχιτεκτονική δομή αυτού του πολυετούς χρηματοδοτικού πλαισίου επαναλαμβάνω, στηρίζεται σε περισσότερη διαφάνεια αλλά και μία πιο σαφή παρουσίαση των διαφορετικών προγραμμάτων, των αναγκών, περισσότερη ευελιξία και αυτό που αναφερθήκατε για τη μεσοπρόθεσμη αναθεώρηση είναι μεγάλη προτεραιότητα για μας. Υπογραμμίζω λοιπόν ότι η πρόταση κανονισμού προβλέπει την αναθεώρησή της μέσω Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δεσμευθεί έτσι ώστε να υποβάλει στις αρμόδιες για τον προπολογισμό αρχές όλες αυτές τις προτάσεις πολύ σύντομα. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να σας ε, υπενθυμίσω ότι η προθεσμία για την υποβολή προπολογιών είναι 6 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα. Ευχαριστώ όλους για τις συνεισφορές σας και τώρα νομίζω ότι μπορούμε να ολοκληρώσουμε το σημείο αυτό και να περάσουμε στο επόμενο. Πρόκειται για το σημείο 8 της ημερησίας διάταξης. Πρόκειται για την ψηφιακή Ευρώπη για την περίοδο 2021-2027 βάσει του άρθρου 54 του κανονισμού. Η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών είναι 7 Σεπτεμβρίου στις 2. Θα ψηφίσουμε στις 10 Οκτωβρίου εδώ στην Επιτροπή και δεν γνωρίζω ακριβώς πότε η αρμόδια επιτροπή, η Επιτροπή Ήτρε θα καθορίσει την ψηφοφορία. Η Ήτρε έχει πάρει αποφάσεις εξαιρετικά φιλόδοξες, θέτοντας την ψηφοφορία στην 5η Νοεμβρίου, πρώτη ανάγνωση ελπίζουμε να ολοκληρωθεί στην θητεία του παρόντος Κοινοβουλίου. Θα ήθελα λοιπόν να σας υπενθυμίσω ότι μπορείτε να υποβάλλετε τροπολογίες μέχρι τις 7 Σεπτεμβρίου, Παρασκευή 7 Σεπτεμβρίου στις 2. Και δίνω το λόγο στην εισηγητή. Το η ψηφιακή Ευρώπη θέλει να συνοδεύσει τον ψηφιακό μετασχηματισμό στην Ευρώπη υπέρ των πολιτών και των επιχειρήσεων με ένα προπολογισμό 9,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Διακόπτει ο μιλητή. Now it's okay. To jeszcze raz. Λοιπόν, επαναλαμβάνω, το πρόγραμμα Ψηφιακή Ευρώπη έχει μια πρικοδότηση 9,2 δισεκατομμυρίων ευρώ και στόχος του είναι να συμβάλλει στο ψηφιακό μετασχηματισμό της Ευρώπης υπέρ των πολιτών και των επιχειρήσεων. Το πρόγραμμα επικεντρώνεται σε πέντε συγκεκριμένους στόχους. Καταρχήν είναι η προηγμένη υπολογιστική, δεύτερον τεχνητή νοημοσύνη, Τρίτον, ε, η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο. Τέταρτος στόχος ε, που είναι σημαντικός για τη δική μας ε, Επιτροπή, προηγμένες ψηφιακές δεξιότητες και πέμπτον ανάπτυξη τη βέλτιστη χρήση ψηφιακής δυνατότητας και διαλειτουργικότητα. Σε ό,τι αφορά την Επιτροπή Πολιτισμού, οι δικοί μας αρμοδιότητες αφορούν κυρίως τις ψηφιακές δεξιότητες και τις ψηφιακές ικανότητες. Οι εργαζόμενοι στην Ευρώπη θα πρέπει να μπορούν να αποκτούν προηγμένες ε, ψηφιακές δεξιότητες ε, μέσω ε, διάφορων καταρτήσεων και πρακτικών κατά τη διάρκεια της εργασίας. Για το λόγο αυτό θεωρώ ότι είναι σημαντικό να υποστηρίξουμε τον πολιτιστικό τομέα από αυτή τη σκοπιά κυρίως ε, την, τον τρέχον ψηφιακό, τρέχοντα ψηφιακό μετασχηματισμό. Αυτό είναι σημαντικό και για την πολιτιστική κληρονομιά και γι' αυτό ο ρόλος της ψηφιακής Ευρώπης θα είναι θεμελιώδης ε, στο να υποστηρίξει την Ευρωπαϊκή σε ό,τι αφορά τι συνέργειε, πρέπει να εγγυθούμε τι συνέργειε μεταξύ του προγράμματο Ψηφιακή Ευρώπη και όλων των άλλων προγραμμάτων που συμπεριλαμβάνονται στο πολιετέ δημοσιονομικό πλαίσιο. Από τη σκοπιά όμως των φιλόδοξων στόχων της ψηφιακής Ευρώπης θέλω να υπογραμμίσω ότι σημασία να εγγυηθούμε την πρικοδότηση που προβλέπεται, τα κονδύλια που προβλέπονται. Γι' αυτό προτείνω κάποια συγκεκριμένες τροπολογίες στον προϋπολογισμό. Συγκεκριμένα προτείνω αύξηση στον προϋπολογισμό σε ό,τι αφορά τον ειδικό στόχο 4, δηλαδή τις προηγμένες ψηφιακές δεξιότητες και προτείνω μία προοικοδότηση περίπου 830 εκατομμυρίων ευρώ, δηλαδή 9% του συνολικού προϋπολογισμού, καθώς και 700 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή 7,6% του προϋπολογισμού που έχουν προβλεφθεί αρχικά από την Κομισιόν. Αυτές είναι οι βασικές στοιχές της γνωμοδοτησής μου. Φυσικά είμαι ανοιχτό σε οποιαδήποτε πρόταση από την πλευρά των σχεδόν συγητών και ελπίζω να μπορέσουμε να συνεχίσουμε την καλή μας συνεργασία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κύριε Νιάκοφ, έχετε το λόγο ως πρώτος και όδης εισηγητής. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ και τον εισηγητή κύριο Βέντα, διότι έχει εργαστεί υποδειγματικά και αυτό κατέληξε σε μια εξισορροπημένη γνωμοδότηση. Ο εισηγητής δίνει έμφαση στην προστιθέμενη αξία αυτών των νέων προγραμμάτων, τα οποία θα επηρεάσουν θετικά τον πολιτισμό. Μέσω της ψηφιοποίησης θα βελτιωθεί η πρόσβαση στο πολιτισμικό περιεχόμενο. Το πρόγραμμα είναι αρκετά φιλόδοξο και οι στόχοι επίσης. Θεωρώ όμως ότι τα... η χρηματοδότηση θα μπορούσε να γίνει με καλύτερο τρόπο. το 7,5% πηγαίνει στις ψηφιακές τεχνολογίες. Αυτό, για, κατά τη γνώμη μου, δεν αρκεί. Η χρηματοδότηση εδώ θα έπρεπε να ανέρχεται τουλάχιστον στο 12% του συνολικού προϋπολογισμού. Χρειάζεται λοιπόν αύξηση. Δεν πρέπει να παραμελούμε τις επενδύσεις στην ψηφιακή, στις ψηφιακές υποδομές και στην κατάρτιση των πολιτών έτσι ώστε να τις χρησιμοποιήσουν. Πρέπει να επενδύσουμε σε αυτούς. Πάνω από 800.000 ε, Ευρωπαίων πολιτών ε, δεν έχουν καμία ψηφιακή δεξιότητα και υπάρχουν πολύ περισσότεροι οι οποίοι έχουν πολύ περιορισμένες ε, ψηφιακές δεξιότητες. Χρειάζεται λοιπόν να το αναγνωρίσουμε αυτό και να γίνει επίσης ένας διαχωρισμός ανάμεσα στον ορίζοντα 2020 και τα άλλα προγράμματα δεν καθίσταται σαφές από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το πώς θα ε, αποφύγουμε τις επικαλύψεις. Γι' αυτό θα ήθελα να αναφέρετε αυτό στην γνωμοδότηση. Επίσης, δεν είναι σαφές ποια ε, τι κονδύλια θα επενδύσουν τα κράτη-μέλη. Πρέπει σίγουρα να γίνουν επενδύσεις τόσο στις επιχειρήσεις όσο και στους ε, πολίτες, τους τελικούς χρήστες και επίσης να δοθεί έμφαση στην ποιότητα και όχι μόνο στην ποσότητα. Τα ψηφιακά hub καινοτομία πρέπει επίσης να ε, τονιστούν αρκετά. Και αυτά τα κέντρα θα πρέπει να δημιουργηθούν κατά προτεραιότητα και στην Ήπεθρο και στις αεροκατοικημένες περιοχές. Σας ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Μακλάρκιν έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τον κύριο Βέντα για την έκθεσή του, διότι και η δική μας ομάδα στηρίζει την πρόταση της Επιτροπής και θεωρεί ότι τόσο μικρομεσαίες επιχειρήσεις όσο και εργαζόμενοι θα μπορέσουν να επωφεληθούν, να αποκτήσουν νέες δεξιότητες, να γίνουν πιο αποτελεσματικοί. Ε, τα big data, τα μεγάλα δεδομένα είναι πάρα πολύ σημαντικά για την επιτυχία αυτής της μετάβασης. Επίσης, ε, είναι πολύ σημαντικό να αναγνωρίσουμε την αξία του blockchain. Είναι κάτι που έχει τεράστιο δυναμικό και, να, και αυτό συνεπάγεται ότι πρέπει να καταρτήσουμε τους πολίτες με δεξιότητες σε αυτόν τον τομέα. Τώρα, αυτή η στήριξη θα είναι διαθέσιμη σε όλη την Ευρώπη, θα μπορούν να συμμετέχουν όλοι σε αυτό. Αυτό είναι κάτι που δεν είναι σαφές ακόμα. Επίσης, ε, υπάρχει ευθύνη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και για την ε, κατάρτιση σε δεξιότητες. Οι προηγουμένες δεξιότητες ε, θα έπρεπε να ε, λάβουν ελαφρώς υψηλότερη χρηματοδότηση και να δοθεί επίσης έμφαση στην επανακατάρτιση για να δούμε πώς ακριβώς, επίσης να δούμε πώς ακριβώς θα λειτουργήσουν αυτά τα ψηφιακά κέντρα, αυτά τα hubs, τα συνεργάζονται κυρίως με μικρομεσαίες επιχειρήσεις, με φοιτητές, πώς ακριβώς θα αποφασίζεται πού θα γίνουν επενδύσεις και πόσο. Κάτι που επίσης είναι σημαντικό για την Επιτροπή Πολιτισμού είναι πώς ακριβώς θα βελτιωθούν αυτές οι ψηφιακές δεξιότητες μέσω της ε, κατάρτισης ε, στην εργασία, μέσω ε, μαζικών επιγραμμικών μαθημάτων. Αυτό θεωρούμε πως έχει τεράστιο δυναμικό και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και επίσης πρέπει να εξετάσουμε το πώς διδάσκεται η πληροφορική και η τεχνολογία στα σχολεία για να δούμε τι μπορούμε να βελτιώσουμε. Επίσης, είναι πολύ σημαντικό να προσθεθούν οι μικρομισές επιχειρήσεις ως δικαιούχοι, αλλά και οι νεόφυτες επιχειρήσεις και να συμφωνήσουμε ε, να να συμφωνήσουμε στο ότι η ποιότητα έχει σημασία και όχι η ποσότητα όχι τα ποσοστά, αλλά το σύνολο. Επίσης, να πω ότι συμφωνώ με την προσέγγιση του εισηγητή, να βελτιώσει δηλαδή τους ε, δείκτες σε γενικές γραμμές. Όμως, ε, θα ήθελα να κλείσω λέγοντας ότι η ψηφιακή Ευρώπη μπορεί να αποτελέσει ε, το μέσο το οποίο θα επιτύχει αυτήν την μετάβαση και την ψηφιακή στις ψηφιακές δεξιότητες που όλοι επιθυμούμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Μίχελς έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θεωρώ ότι ο εισηγητής έβαλε τα θεμέλια για να συνεχίσουμε τις εργασίες μας. Είναι πολύ σωστά θεμέλια και θα ήθελα λοιπόν να σας συγχαρώ άλλη μία φορά για το ότι τονίσατε την ενίσχυση του ε, τομέα 4, ε, τις ψηφιακές δηλαδή δεξιότητες. Νομίζω πως... Ε, στην Επιτροπή Πολιτισμού οι ψηφιακές δεξιότητες είναι αυτό που μας απασχολεί περισσότερο. Επίσης, θα, θα πρέπει να φροντίσουμε τη δημιουργία συνεργειών, αλλά να αναγνωρίσουμε ότι υπάρχει υποχρηματοδότηση. Να μου το πείτε παρακαλώ, διακόπτη από το Προεδρείο. Εντάξει τώρα. Ναι, μπορείτε να ξεκινήσετε από την αρχή. Νομίζω πως ε, δεν κατάλαβα καλά ο εισηγητής. Ναι, θα αρχίσω από την αρχή, τέλος πάντων. Θεωρώ λοιπόν πως η πρότασή του είναι πάρα πολύ καλή. Χαιρετίζουμε ιδιαίτερα την αύξηση που προτείνει ο εισηγητής. Ιδιαίτερα στον ε, στόχο αριθμό 4, τις ψηφιακές ε, δεξιότητες. Διότι γνωρίζουμε όλοι ότι εάν ε, θέλουμε να δημιουργήσουμε συνέργειες ε, θα πρέπει να αναγνωρίσουμε επίσης και την ε, χρόνια υποχρηματοδότηση των project αυτών. Επίσης, όπως είπατε κι εσείς, στην τροπολογία 32 πρέπει να αναγνωρίσουμε τη στήριξη στους ε, πολίτες της Ευρώπης, στην ε, διευκόλυνση της πρόσβασης στα πολιτισμικά αγαθά μέσω της ε, ψηφιακής τεχνολογίας, μέσω Wi-Fi ας πούμε. Αυτό βέβαια δεν είναι τίποτα μπροστά στο σύνολο, όμως νομίζω πως σε θέματα χρηματοδότηση έχουμε μάθει να μην ζητάμε πολλά. Επίσης, η κατάρτιση, η επανακατάρτιση που προτείνεται ε, ε, αναφέρομαι στις τροπολογίες 12 ε, και 13. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, πιστεύουμε, να διασφαλίζεται η επανακατάρτιση, επανεκπαίδευση. Όμως πρέπει να είμαστε πιο συγκεκριμένοι και όχι τόσο γενικοί. Μετά, Έχουμε και κάποιες δικές μας προτάσεις διεύρυνσης του πεδίου Από τη μία γνωρίζουμε ότι η πολυγλωσία είναι ωφέλιμη για την εσωτερική αγορά. Από την άλλη όμως βλέπουμε ότι υπάρχουν ορισμένες γλώσσες που υπερτερούν και υπερέχουν ε, σε ορισμένους τομείς. Για παράδειγμα, στην πληροφορική χρησιμοποιούν όλοι λίγο πολύ μία γλώσσα. Χρειάζεται λοιπόν να αναγνωρίσουμε ότι πρέπει να δώσουμε περισσότερες ευκαιρίες ε, στην ε, πολυγλωσσία και να δώσουμε έμφαση στην μετάφραση κειμένων σχετικών με αυτές τις τεχνολογίες. Μετά, το σημείο όπου τονίζεται η διαλειτουργικότητα. Να πω ότι το καλωσορίζω μεν, αλλά με κάποιο δισταγμό, διότι όλοι οι πολιτικοί το ζητούν, από την άλλη όμως υπάρχει δισταγμό στη χρηματοδότηση, ε, δεν θέλουν να δώσουν δημόσια κονδύλια, αλλά για μας αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και αν όταν μάλλον καταθέσουμε τροπολογίε, θα ήθελα να πάμε και προ αυτήν την κατεύθυνση. Αυτά από μένα προ το παρόν. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ για την συνεργασία. Κυρία Τρίπελ, τελευταία σκιώδη. Ευχαριστώ, θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή, τον κύριο Βέντα. Και θα απαντήσω πρώτα στου δύο τελευταίους ομιλητές. Ναι, Σίγουρα είναι πάρα πολύ σημαντικέ οι μικρομεσαίε επιχειρήσει, ιδιαίτερα γιατί υπάρχει αυτή τη στιγμή η μονοπωλιακή αυτή δομή των μεγάλων επιχειρήσεων των ΚΑΠΑ. Γι' αυτό και θα πρέπει να στηρίξουμε μια ιδιαίτερη προσέγγιση και αυτό είναι και τελικά και ο στόχος αυτού του προγράμματος να στηρίξουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Συμφωνώ απολύτως. Όσον αφορά τα χάπης καινοτομία ε, για την ψηφιακή οικονομία, ναι, είναι πάρα πολύ επίγον να αναπτύξουμε μία νέα πολιτική στον τομέα του ανταγωνισμού. Υπάρχουν όμως πάρα πολλές αντιφάσεις. Ήταν ε, την τελευταία δεκαετία μόδα να παρέχουν όλα τα πανεπιστήμια online μαθήματα. Τελικά όμως ε, αυτό που σήμερα γνωρίζουμε είναι ότι οι περισσότεροι φοιτητές ζητούν ε, ένα μείγμα, αν θέλετε, παραδοσιακών ε, μαθημάτων με έναν καθηγητή στον οποίο μπορούν να απευθυνθούν, να μιλήσουν, να ανταλλάξουν και βεβαίως τα μαθήματα online. Κυρία Μίχελς. Βεβαίως είναι καθοριστικό το πρόγραμμα Media. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το να δημιουργήσουμε νέες δεξιότητες στις νέες τεχνολογίες, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης οι νέοι αλλά και οι λιγότερο νέοι θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να αποφασίσουν ποια είναι η ποιότητα, αν θέλετε, του περιεχομένου που τους προσφέρεται. Αλλιώς, αν δεν μπορούμε να κρίνουμε, αν δεν μπορούμε να συγκρίνουμε και να αποφασίσουμε, γνωρίζοντας το περιεχόμενο, νομίζω ότι μπορούμε να μιλήσουμε για αναλφαβητισμό. Ναι, ε, όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Βεβαίως εδώ προκύπτει και το θέμα των πνευματικών δικαιωμάτων, αλλά θα πρέπει να είμαστε σε δυνατότητα να χρηματοδοτήσουμε και να μετατρέψουμε όλο αυτό το περιεχόμενο σε ψηφιακό. Και βάσει κανόνων, ακριβώς όπως κάνουμε τώρα με το copyright, με τα πνευματικά δικαιώματα. Οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις παίζουν πρωταεργικό, ηγετικό ρόλο σε θέματα γλωσσικά, στους ε, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, τις νέες τεχνολογίες και αυτό είναι κάτι που σίγουρα θα πρέπει να το στηρίξουμε. Είναι τμήμα του Εράσμους και του Horizon. Και τώρα θα κάνω τις γενικές μου παρατηρήσεις για την ψηφιακή Ευρώπη. Βρισκόμαστε εν μέσω τα τελευταία 20 χρόνια μιας επανάστασης τεχνολογικής η ψηφιακή επανάσταση είναι πραγματικότητα, γι' αυτό και πρέπει να μιλήσουμε για ανταγωνισμό. Οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις δεν παίζουν πρωταρχικό ρόλο εδώ. Έχουμε πρόβλημα και με την Κίνα και με τις Ηνωμένε Πολιτείε. και θα πρέπει να βιαστούμε, να τους προλάβουμε. Χρειαζόμαστε κανόνες, χρειαζόμαστε όμως και δεξιότητες οι δεξιότητες δεν είναι απλώς θέμα τεχνολογίας, προγραμματισμού, χρήσης εξοπλισμών. Είναι και θέμα κρίσης. Ποια είναι τα συν και τα πλήν της τεχνητής νομιμοσύνης, παραδείγματος χάρη. Στηρίζουμε την τεχνική νομιμοσύνη και φυσικά καθημερινά διαβάζουμε στον τύπο τις νέες προκλήσεις που θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε, ακριβώς επειδή εξελίσσεται και προοδεύει η τεχνητή νοημοσύνη και όλοι οι τομείς ε, που σήμερα στην Ευρώπη δυστυχώς δεν είναι πρωτοπορία. Θα ήθελα να συζητήσουμε μια βασική αντίφαση. Μιλούμε για την ενιαία ψηφιακή αγορά. Θέλουμε να στηρίξουμε και να προωθήσουμε την ψηφιακή Ευρώπη. Δεν υπάρχει όμως ε, ενιαία ψηφιακή αγορά. Γιατί? Γιατί θέλουμε να υπάρχει γλωσσική και πολιτιστική πολυμορφία. Και αυτό συνδέεται άμεσα με την γεωγραφία της Ευρώπης. Δεν έχουμε μία γλώσσα, δεν έχουμε ένα πολιτισμό. Και αυτό ισχύει για τη μουσική, για τον κινηματογράφο και για τη λογοτεχνία. Γι' αυτό και θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί από τη μία να τηρούμε και να σεβόμαστε την πολιτιστική γλωσσική πολυμορφία. Γι' αυτό και η μεταρρύθμιση στον τομέα των πνευματικών δικαιωμάτων, το ευρωπαϊκό copyright θα πρέπει να αποτελέσει κεντρική ιδέα της πολιτικής μας. Αυτό πρέπει να είναι στην καρδιά, αν θέλετε, της οικοδόμησης αυτού που θέλουμε να δημιουργήσουμε σαν ενιαία ψηφιακή αγορά. Δεν είμαστε Κίνα, δεν είμαστε Ηνωμένε Πολιτείε, γι' αυτό και η ψηφιακή Ευρώπη θα πρέπει να καθοριστεί βάσει της δικής μας προσέγγισης. Είμαστε η Επιτροπή Πολιτισμού, δεν είμαστε Ήτρε. Μην ξεχνάμε λοιπόν ότι υπάρχουν αντιφάσεις μεταξύ των στόχων, μεταξύ της αγοράς, μεταξύ της οικονομίας και της πολιτικής στικής πολυμορφίας. Δεν είμαι κατά της καινοτομίας, δεν είμαι κατά της τεχνολογίας, αλλά πρέπει να βρούμε μοντέλα που να ανταποκρίνονται στο ποιοτικό περιεχόμενο του πολιτισμού που θέλουμε να στηρίξουμε. Θα σε ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Να δώσω τώρα το λόγο στην κυρία Κώστα. Κάποια σχόλια Εκτιμώ το κείμενο του συναδέλφου. Νομίζω ότι είναι καλό. Θα πρέπει όμως ε, να ζητήσουμε συνέργειες μεταξύ των πέντε στόχων της ε, στρατηγικής ψηφιακή Ευρώπη, κυρίως ό,τι αφορά τις ε, προηγουμένες αρμοδιότητες, τις προηγουμένες δεξιότητες και πιστεύω ότι θα πρέπει να υπάρχει και μία αναφορά στο να υποστηρίξουμε την ψηφιοποίηση όχι μόνο της, ε, των δημιουργικών ε, και πολιτιστικών βιομηχανιών, αλλά να δημιουργήσουμε και μια συνέργεια μεταξύ ψηφιοποίησης, πολιτιστικής κληρονομιάς και έρευνας έχουμε νέες μορφές επικοινωνίας ε, και είναι κλειδί έρευνα. από τα νέα ψηφιακά μουσεία, παραδείγματος χάρη, μέχρι ε, και την δυνατότητα μεγαλύτερης πρόσβασης ε, μέσω της γλώσσας παραδείγματος χάρη μπορεί κάποιοι νέοι, τα παιδιά να έρθουν πιο κοντά στον ευρωπαϊκό πολιτισμό ε, θα πρέπει λοιπόν να δημιουργήσουμε ένα τομέα που να ξεκινά από την πολιτιστική κληρονομιά και να φτάνει μέχρι τις καινοτόμε επιχειρήσεις και υπηρεσίες. Έτσι λοιπόν θα πρέπει αυτά να τα βάλουμε δίπλα-δίπλα. Νομίζω ότι ο προϋπολογισμός είναι πολύ μειωμένος, πολύ χαμηλός, όπως είπε και ο συνάδελφος Νέκοφ. Χρειάζεται δηλαδή μεγαλύτερη αύξηση του προπολογισμού, μεγαλύτερη και που ζήτησε ο εισηγητής. Και θέλω να αναφερθώ και σε αυτό που συζητήσαμε πριν. Στην επένδυση που θα κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην παραγωγή ψηφιακού περιεχομένου. Εμείς έχουμε και τη φιλοδοξία να παράγουμε τέτοια περιεχόμενα. Δεν ε, θέλουμε μόνο να μιλάμε για ψηφιοποίηση, αλλά θέλουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί σε παγκόσμιο επίπεδο σε ό,τι αφορά τα ψηφιακά περιεχόμενα. Και σε ό,τι αφορά τώρα την εκπαίδευση, νομίζω ότι πρέπει να επενδύσουμε περισσότερα σε αυτό που αποκαλούμε MOOC, δηλαδή ε, στην ψηφιακή διδακτική, ε, όχι μόνο με την εξαποστάσεως εκπαίδευση, αλλά και με blended συστήματα. Ο εισηγητής πολύ σωστά αναφέρεται ε, στην απέτηση να έχουμε κατεξουσιοδότηση πράξης, γιατί είναι ένα σενάριο που είναι υπό τροποποίηση ίσως θα πρέπει να έχουμε μία γενική γραμμή. Το λέω και εγώ για τον εαυτό μου ε, ως εισηγήτρια για την Δημιουργική Ευρώπη. Δηλαδή, πρέπει να δούμε ποια είναι η στρατηγική που θέλει να έχει το Κοινοβούλιο προ αυτή την κατεύθυνση. Γιατί αν εμεί θεωρούμε ότι στα 7 χρόνια αλλάζει πάρα πολύ γρήγορα το σενάριο και το γνωρίζουμε και το Κοινοβούλιο ουσιαστικά ε, αν θέλει να κάνει μια νέα, ένα νέο επαναπροσδιορισμό των πολιτικών ε, στο χρόνο πρέπει να αποφασίσουμε ποια στρατηγική θέλουμε. Είδαμε τι συζητήσαμε και στην ε, έκθεση της ε, κυρίας ε, Κάμερβερτ. Δηλαδή ζητήθηκε εκεί μια ενδιάμεση αναθεώρηση υποχρεωτική Ω προ τον επαναπροσδιορισμό των πολιτικών. Θα ακολουθήσουμε αυτή την κατεύθυνση ή θα έχουμε κατεξουσιοδότηση πράξη γενικά. Γιατί αυτό ουσιαστικά αφορά με οριζόντιο τρόπο όλα τα προγράμματα. Αυτό θα πρέπει να το αποφασίσουμε πολιτικά και ως ομάδες. Γιατί νομίζω ότι πρέπει να δώσουμε μια εναρμονισμένη απάντηση. Επίσης, δεν μου φαίνεται ακόμα ικανοποιητικός ε, στο κείμενο της ε, Κομισιόν ο τρόπος που θα καταστούν διαλειτουργικά τα ευρωπαϊκά προγράμματα. Εδώ πάντοτε μιλάμε για κάτι ευκταίο. Δηλαδή τα προγράμματα θα πρέπει το ένα αμοιβαία να παραπέμπει στο άλλο. Εμείς πρέπει να δούμε πώς θα γίνει αυτή η διάρθρωση. Αυτό μας λείπει ακόμα και είναι ένα γενικό θέμα που θα πρέπει να συζητήσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Εξ ονόματος της Επιτροπής θέλει κάποιος να πάρει το λόγο. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Ειλικρινά ευχαριστούμε για την εξαιρετική αυτή έκθεση του εισηγητή αλλά και των σκιωδών καθώς και για τη στήριξη όλης της Επιτροπής στα θέματα αυτά, τις ψηφιακές δεξιότητες, το πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη και τον πολιτισμό. Νομίζω ότι μοιραζόμαστε τους ίδιους στόχους και την ίδια φιλοδοξία. Θα σας δώσω κάποιες επιπλέον ε, πληροφορίες και στοιχεία που ουσιαστικά αφορούν όλες τις προτάσεις μας και τις ψηφιακές δεκτυότητες όπως επεριέχονται στο πολιετές δημοσιονομικό αυτό πρόγραμμα. Αντιμετωπίζουμε δυσκολίες στον τομέα αυτό στην Ευρώπη από τις πρώτες βαθμίδες της εκπαίδευσης στο Δημοτικό Σχολείο μέχρι και τις πανεπιστημιακές και ακαδημαϊκές σπουδές. Γι' αυτό και στο πολιετές αυτό πρόγραμμα θέλουμε να στοχεύσουμε τις δεξιότητες, αλλά και την στήριξη την οικονομική για να μπορέσουμε να τις ε, παρέχουμε σε όλα αυτά τα επίπεδα. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω πώς ακριβώς σχεδιάσαμε αυτό το πρόγραμμα. Ξεκινήσαμε με το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το ESF, Μέσω των επιχειρησιακών προγραμμάτων τα κράτη-μέλη έχουν θέσει προτεραιότητες. Έχουν θέσει δύο πολύ σημαντικές προτεραιότητες για τις ε, ψηφιακές δεξιότητες και τη στήριξή τους. Και όσον αφορά την υλοποίηση αυτών των πρώτων φάσεων, τα διαρθρωτικά ταμεία μπορούν σήμερα να επαναπροσδιορίσουν προτεραιότητες έτσι ώστε να στηρίξουν αυτές τις πρωτοβουλίες. 200 εκατομμύρια ετήσιο ποσό διατίθεται, καθώς και υποχρεωτικά προγράμματα για τις περιπτώσεις απολυμένων εργαζομένων οι οποίοι θέλουν να επανεσωματωθούν στην ε, αγορά εργασίας. Επίσης υπάρχουν ε, οργανώσεις σεμιναρίων μαθημάτων ε, στα πλαίσια της ε, επαγγελματικής κατάρτισης. Έχουμε το Horizon Europe, δίνονται υποτροφίες ε, για μεταπτυχιακά, για διδακτορικά, χρηματοδοτούνται προγράμματα κατάρτισης βάσει των προγραμμάτων Marie Curie και θέλουμε να στηρίξουμε κάθε είδους ε, δεξιότητες στον ψηφιακό τομέα από τα πρώτα επίπεδα μέχρι και τα εξαιρετικά προηγμένα. Παρακολουθώντας ε, τις νεότερες εξελίξεις στην ε, τεχνολογία, στην έρευνα, στηρίζοντας κοινά ερευνητικά κέντρα και προγράμματα. Γι' αυτό και βλέπετε ότι όλες αυτές οι συνεργασίες που μπορούν και θα αναπτυχθούν είναι σε πολλά διαφορετικά επίπεδα. Για το Ευρωπαϊκά, πολλοί από εσά αναφέρθηκαν και φαίνεται να δείχνετε ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Το Ευρωπαϊκά Ζητώ συγγνώμη, δεν έχω τις σημειώσεις μου εδώ. Τέλος Απριλίου έγινε μια αξιολόγηση και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ουσιαστικά υιοθέτησε μια νέα στρατηγική για το Ευρωπαϊκό μετά από μια ανεξάρτητη αξιολόγηση. Η έκθεση αυτής της ανεξάρτητης αξιολόγησης θα δημοσιευθεί τις επόμενες εβδομάδες και μετά το 2020 θα ακολουθήσουμε τα πορίσματα της έκθεσης αυτής με μια επιπλέον χρηματοδότηση της τάξης των 20 εκατομμυρίων ευρώ οι δράσεις για να προωθήσουμε τις ψηφιακές δεξιότητες όπως ξέρετε υπάρχουν ήδη τα κέντρα στο διαδίκτυο, οι πλατφόρμες και αυτό σε πανευρωπαϊκό επίπεδο με συγκεκριμένα κέντρα, με ενημερωτικές καμπάνιες για να μειωθεί ο ψηφιακός αναλφαβητισμός και αυτό βεβαίως ενσωματώνεται και σε πολλές άλλες οδηγίες όπως την προστασία των παιδιών και όλες τις οδηγίες οι οποίες αναφέρονται στα πολυμέσα και στο διαδίκτυο και τα παιδιά. Σας ευχαριστώ πολύ και θα σας ενημερώσουμε όσο εξελίσσεται η προσπάθειά μας. Ευχαριστώ πολύ κυρία Κώστα. Πολύ σύντομα. Κάτι να διευκρινίσω μόνο. Υπόθηκε ότι δεν υπάρχει καμία ειδική αναφορά στο Εράσμους. Θέλω να επενθυμίσω ότι δεν αναφέρθηκε η e-student card εδώ και καιρό θα έπρεπε η ε, Κομισιόν να έχει συνεργαστεί με τη ΓΑΜΑ Connect γιατί πρόκειται για ένα σημαντικό εργαλείο που έχει προβλεφθεί ήδη και στην διάστηση του Γκέντεμπορκ ως προτεραιότητα από τους υπουργού Παιδείας, που δίνει τη δυνατότητα στους νέους Ευρωπαίους φοιτητές να μπορούν όχι μόνο να έχουν μία κάρτα, όπου θα αναγράφονται όλες τους οι αλλά θα μπορούν να έχουν και πρόσβαση σε όλη την Ευρώπη, ε, σε διάφορες ε, εκδηλώσεις ε, πολιτιστικές. Είχα από τη ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑ παιδείας και τη ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑ Κοντέκτ ότι είχε προχωρήσει αυτό το σχέδιο για να καταστεί λειτουργική η κάρτα για το 2021. Όμως ε, δεν είδα κανέναν ε, να αναφέρεται σε αυτό το πρόγραμμα για ε, συγγνώμη που ξέχασα να το αναφέρω πριν. Ευχαριστώ. Και τώρα να δώσω το λόγο στον κύριο Βέντα για, τρία, για τα τρία λεπτά για τα τελικά σχόλια. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους για τα σχόλια. Όλες ε, αυτές οι παρατηρήσεις μας δείχνουν πόσο σημαντικό είναι αυτό το πρόγραμμα για όλους μας. Ε, όπως είχα πει στην αρχικά μου σχόλια, θέλουμε καταρχήν να εγγυηθούμε τα κονδύλια που προβλέπονται για το πρόγραμμα αυτό και κατόπιν όλων αυτών ε, των ε, σχολείων αναμένω και τις τροπολογίες από τους συναδέλφους, όμως υπενθυμίζω ότι δεν έχουμε πολύ χρόνο στη διάθεσή μας. Επομένως, θα ήθελα να ζητήσω κάποια κατανόηση από όλους και σας καλώ να παρουσιάσετε τις πιο σημαντικές ε, τροπολογίες. Αυτές που θεωρείτε πιο σημαντικές για τους συντάκτες αλλά και για την Επιτροπή Πολιτισμού αναφέρθηκε στο ότι λείπουν δεξιότητες σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ακόμη και σε επίπεδο δημοτικού. Έχουμε έλλειψη σε ψηφιακές δεξιότητες, όμως θα πρέπει να αναπτυχθούν αυτές πολύ γρήγορα, γιατί έχουμε πολύ μεγάλες εξελίξεις σε αυτό τον τομέα. Έτσι λοιπόν απευθύνω έκκληση στους συναδέλφους να είναι ευέλικτοι έτσι ώστε να μπορέσουν πολύ σύντομα να παρουσιάσουν αξιόλογες τροπολογίες και θέλω να επενθυμίσω ότι η Επιτροπή είναι αυτή που τελικά ε, είναι καθήλυνα αρμόδια. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ για όλες τις ε, συνεισφορές σας. Ευχαριστούμε τα μέλη της Επιτροπής μας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τον εισηγητή για την εργασία του. Ολοκληρώνουμε λοιπόν αυτό το σημείο στην ουρήση διάταξη και περνάμε τώρα στο σημείο 9, πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του προγράμματο πλαισίου Έρευνα και κοινοτομία ορίζων Ευρώπη και των κανόνων συμμετοχή και διαδοσή του. Ο κύριο Λουίτζι Μοργκάνο είναι ο εισηγητής 5 ε, Σεπτεμβρίου στι 2 το μεσημέρι. Είναι η προθεσμία κατάθεση τροπολογιών και θα ψηφίσουμε στι 10 Οκτωβρίου. Και η συνδεδεμένη επιτροπή, η Ήτρε, θα ψηφίσει στις 21 Νοεμβρίου. Δίνω αμέσω το λόγο στον κύριο μόργκανο για πέντε λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα έλεγα ότι είναι στενό το χρονοδιάγραμμα και ε, επομένως εγώ από την πλευρά μου θα προβώ στην παρουσίαση αυτής ε, της ε, γνωμοδότησης και η γνωμοδότηση για το νέο πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα και την καινοτομία για την περίοδο 2021-2027, ορίζον Ευρώπης, ξέρετε, ότι έχει ένα πολύ στενό χρονοδιάγραμμα. Ε, ουσιαστικά ε, ε έπρεπε να εγκαταλείψω την δική μας γνωμοδότηση. Ε, βέβαια δεν είναι κάτι αποδεκτό. Θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Στεφανή Μπιασόλη από τη Γραμματεία της Επιτροπής και τους βοηθούς μου. Όπως ε, θα έχετε διαβάσει ήδη στο σχέδιο γνωμοδότησης, σε όσα μπόρεσαν να γίνουν μέσα στο λίγο χρόνο, προσπάθησα να παρουσιάσω κάποιες από τις κύριες πολιτικές προτεραιότητες της Επιτροπής μας γνωρίζοντας ότι σίγουρα θα χρειαστεί να παρουσιαστούν και περαιτέρω τροπολογίες για να συμπληρωθεί ε, το κείμενο αλλά και για να διευκρινιστεί υπό το φως των πληροφοριών που έχουν συλλεχθεί κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών διακοπών. Θα ήθελα λοιπόν να υπογραμμίσω τα εξή. Αφενό, να γνωρίζω την προσπάθεια από την πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή που έχει προβλέψει μια αύξηση του προπολογισμού σε σχέση με το προηγούμενο πρόγραμμα, φτάνοντα στα 94 δισεκατομμύρια και 100 εκατομμύρια ευρώ. Θεωρώ όμως ότι ε, τα συνολικά κονδύλια, η συνολική πρικοδότηση για αυτό το πρόγραμμα Ναυαρχίδα δεν ε, είναι επαρκώς φιλόδοξη, λαμβάνοντας υπόψη τους στόχους που έχουν προταθεί. Έτσι λοιπόν έχω προτείνει στο κείμενο να αυξήσουμε τη χρηματοδότηση τουλάχιστον στα 120 δισεκατομμύρια. Επίσης, λαμβάνοντας ε, υπόψη την πολιτική συμφωνία που επιτεύχθη στην Ήτρε μεταξύ των εισηγητών Νίκα και Έλερ, από τους οποίους ε, έμαθα ε, στη συνέχεια, μπορώ να σας πω ότι η δική μου πρόθεση είναι να προσανατολιστώ προς τα πάνω ε, και να προτείνω μια τροπολογία έτσι ώστε να περάσουμε από τρέχουσες τιμές σε σταθερές τιμές για να μπορέσουμε να βασιστούμε σε ένα συγκεκριμένο αριθμό ανεξάρτητα από το πληθωρισμό. Δεύτερον, είναι απαραίτητο να υποστηρίξουμε σε μεγάλο βαθμό τον πρώτο πυλώνα ανοιχτή επιστήμη. Και εδώ Αναφέρομαι συγκεκριμένα στις ε, δράσεις ε, που έχουν να κάνουν ε, με το πρόγραμμα Μαρκιουρί. Τώρα, κατόπιν των πληροφοριών που έλαβα αυτή την τελευταία περίοδο, μπορώ να σας πω ότι θα παρουσιάσω τροπολογίες για να ζητήσω τουλάχιστον 11 δισεκατομμύρια ευρώ και 3.300 εκατομμύρια για τις υποδομές έρευνας. Σε πραγματι μιας, ε, ενός πραγματικού ευρωπαϊκού χώρου έρευνας που να προβλέπει καλύτερη σύνδεση μεταξύ έρευνας, ε, επιστημονικής αρισίας, καινοτομία και πανεπιστημίων θα πρέπει να είναι στο επίκεντρο του προγράμματος Horizon Ευρώπης και να διέπει όλους τους πυλώνες. Τώρα, σε σχέση με το δεύτερο πυλώνα, προκλήσει σε παγκόσμιο επίπεδο και βιομηχανική ανταγωνιστικότητα, αυτό είναι ο τίτλο, ε, δεν μπορούμε παρά με ικανοποίηση να σημειώσουμε ότι ιδίω ο πόλο, ο θεματικό, ε, συμμετοχική και ασφαλή κοινωνία, έχει αναγνωριστεί ότι παίζει σημαντικό ρόλο και η ευρωπαϊκή πολιτιστική κληρονομιά. Και βάσει μια εις καλοκαιρινή ανάλυσης, οι αυγουστιάτικες αν θέλετε, θεωρώ ότι ε, η πτυχή της ασφάλειας θα πρέπει να διαχωριστεί από τα υπόλοιπα. Έχουμε μια ακόμη πιο γενική συζήτηση που θα μπορούσε να γίνει λοιπόν. Ε, σε αυτό το κλάστερ πάντως χρειάζεται να βάλουμε νέους ε, τομείς παρέμβασης. Θεωρώ ότι θα έπρεπε να ε, τονίσουμε περισσότερο τον πολιτισμό και το στρατηγικό ρόλο του πολιτιστικού και δημιουργικού τομέα για να ε, μπορέσουμε να υλοποιήσουμε μια δημιουργική και μορφωμένη κοινωνία ε, και μια ακόμη πιο συμμετοχική κοινωνία. Έτσι λοιπόν έχω κάνει ρητή αναφορά στη στρατηγική δυναμική της ε, πολιτιστικής και δημιουργικής βιομηχανίας ακόμη και στο πλαίσιο της ψηφιακής καινοτομίας λαμβάνοντας υπόψη τον διτό χαρακτήρα, δηλαδή ότι προωθεί την οικονομική ανάπτυξη και προστατεύει την πολιτιστική και γλωσσική πολυμορφία κτηνοτροφία στην Ευρώπη. Έχοντα λοιπόν υπόψη αυτού του νέου τομεί παρέμβαση που θα διευκρινίσω και εγώ στι τροπολογίε μου που θα τι θέσω βέβαια και υπόψη των σχεδόν συγκητών για να μπορέσουν να τι αξιολογήσουν και το ταχύτερο να φτάσουμε σε πραγματική σύγκληση. Πιστε, έχω κατά νου και τα 5G, ε, τη διαχείριση του copyright και θα ζητήσω να αυξηθεί ο προπολογισμό για αυτό το θεματικό πόλο και να πάμε τουλάχιστον στα 3,3 δις. Έτσι λοιπόν, ε, φυσικά οι προτάσεις αφορούν ακριβώς την ε, συγκεκριμένη παρέμβαση σε συγκεκριμένους ε, τομείς των κεφαλαίων η τεχνολογική καινοτομία όπως το ίντερνετ των πραγμάτων, ε, οι ε, τεχνολογίες παροχής βοήθειας ε, που εφαρμόζονται ήδη σε ένα αρχαιολογικό χώρο ή σε ένα βιβλίο μπορούν να διευκολύνουν την πρόσβαση στον πολιτισμό και στη δημιουργικότητα, συνεισφέροντας συγκεκριμένα στην υλοποίηση της πλήρους ένταξης των ατόμων αυτών σήμερα. Δεν ξέρουμε βέβαια που θα φτάσουμε τα επόμενα 10 χρόνια που καλύπτει το πρόγραμμα αυτό. Ήδη ε, εργαζόμαστε στην δυνατότητα να καταστήσουμε ορατές τις εικόνες ε, σε ανθρώπους με προβλήματα όρασης, ε, μεταμορφώνοντάς τις σε τριδιάστατες εικόνες. Επίσης, πρέπει να χάρη έχουμε τεχνολογίες ε, που ε, διευκολύνουν την πρόσβαση σε ανθρώπους με γνωστικές ε, δυσκολίες. Πρέπει να χάρη έχουμε νεολογικούς χάρτες για τους δυσλεξικούς προκειμένου να συνεισφέρω στην ανάλυση και στην εξέβρεση λύσεων για την αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων που αντιμετωπίζει η Ευρώπη, ως παραδείγματος χάρη του μεταναστευτικού φαινομένου. Ε, το, πρόγραμμα, το πρόγραμμα αυτό ε, θα έπρεπε επίσης να υποστηρίξει την ε, έρευνα στις ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες και βασική έρευνα αλλά και εφαρμοσμένη έρευνα. Τέλος, σε σχέση με την δυνατότητα να προσφύγουμε σε συνέργειες μεταξύ επιστήμης, τεχνολογίας, πολιτισμού και τεχνών για να έχουμε μία ε, βιώσιμη και ποιοτική καινοτομία, θεώρησα σημαντικό να συμπεριλάβω και την δημιουργική Ευρώπη που δεν είχε προβλεφθεί στον κατάλογο των πιθανών προγραμμάτων της Ένωσης με την οποία ε, μπορεί να ε, έχει διαδραστική επίδραση το ορίζον Ευρώπης. Και κλείσω, είμαι βέβαιος ότι μαζί με τη συνεισφορά των σκιωδών συγητών ε, και όχι μόνο θα μπορέσουμε να παρουσιάσουμε στην Επιτροπή Ήτρε που είναι η καθήλια αρμόδια επιτροπή μια διαρθρωμένη και συνεκτική γνωμοδότηση που να λάβει υπόψη όλες τις πολιτικές προτεραιότητες της δικής μας Επιτροπής. Και ελπίζουμε να μπορέσει να καταστεί ε, μέρος αυτού του νέου εμβληματικού προγράμματος της Ευρώπης, το οποίο στόχος είναι η ενίσχυση τη επιστημονικής και τεχνολογική βάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προωθώντα και περασπίζοντας την ενεργητική δραστηριότητα και την καινοτομία που θα μας οδηγήσουν σε μια βιώσιμη ανάπτυξη και σε βιομηχανική ανταγωνιστικότητα προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής εκατομμυρίων πολιτών. Επίσης είμαι επιπισμένος ότι όπως κάναμε και στο παρελθόν έχουμε πραγματικούς λόγους να υποστηρίξουμε κάποια πράγματα να ληφθούν υπόψη δεόντως και να ενταχθούν σε αυτόν τον κανονισμό. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ τον εισηγητή. Είμαι και εγώ σκιώδης του ΕΛΚ, γι' αυτό θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας τις απόψεις μου αμέσως και μετά θα δώσω το λόγο στους υπόλοιπους σκιώδης εισηγητές. Ε, θεωρώ λοιπόν πως ε, είναι πολύ θετικό ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αύξησε αυτή τη γραμμή του προπολογισμού από 31 σε 69 εκατομμύρια. Το έχουμε ακούσει πολλές φορές, ε, πρέπει να προσανατολίσουμε τις επενδύσεις μας στο μέλλον και είμαι σίγουρη ότι οι επόμενες γενιές ε, θα έχουν καλύτερο επίπεδο διαβίωσης με αυτόν τον τρόπο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να γίνει λόγος για την έρευνα και την καινοτομία και να τονίσουμε επίσης ότι για εμάς την Επιτροπή Πολιτισμού και ε, εκπαίδευσης ε, είναι σημαντικό να επικεντρωθούμε κυρίως ε, στην πολιτισμική διάσταση, ενώ η Επιτροπή ΉΤΡΕ στην βιομηχανική. Οι υποδομές και καινοτομία πρέπει να βελτιωθούν και να δημιουργηθούν επίσης, διότι αν δεν υπάρχει κατάλληλη υποδομή, δεν θα μπορέσουμε να επιτύχουμε την πρόοδο που επιθυμούμε. Δεν θα μπορέσει να λάβει χώρα η ψηφιοποίηση. Δεν θα μπορέσουμε να προστατεύσουμε τις ε, πολιτισμικές μας αξίες. Θεωρώ για αυτούς τους λόγους σημαντικό το να έχουμε τη συμμετοχή όλων. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να τονίσουμε την συμμετοχή στην εκπαίδευση και θα ήθελα να ζητήσω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να στηρίξει τα προγράμματα έβρεσης ε, αξιόλογων ε, ταλέντων, να μην τα παραμελεί. Χρειαζόμαστε ταλαντούχους ανθρώπους ε, για να καταφέρουμε όλα αυτά. Και αυτό, ξέρετε, ξεκινά από την παιδική ηλικία. Όταν ε, ανακαλύπτουμε κάποιο ταλέντο πρέπει να το στηρίζουμε, να το προωθούμε. Μόνο έτσι θα επιτύχουμε την αριστεία. Εάν αναγνωρίζουμε και στηρίζουμε τα ταλέντα για όλη τη ζωή. Θα ήθελα λοιπόν ε, να καταθέσω μια σχετική τροπολογία που θα τονίζει το σημείο αυτό. Και κάτι άλλο. Ε, σε ό,τι αφορά το ότι ο πολιτισμός και η δημιουργικότητα δεν τονίζονται επαρκώς στην δομοδότηση, να το προσυπογράψω κι εγώ. Υπάρχει μία διαφορά ανάμεσα στα ε, παλιά κρατημέλη και στα νέα κρατημέλη. Δεν υπάρχει δίκαιη κατανομή της χρηματοδότησης. Τα δύο τρίτα της χρηματοδότησης πηγαίνουν στα παλιά κρατημέλη. Και στο πλαίσιο ε, αυτό λοιπόν βρίσκουμε να γέρνει η πλάστικα υπέρ των ε, παλαιών κρατών μελών. Χρειάζεται λοιπόν αυτό να αλλάξει. Γι' αυτούς τους λόγους θεωρώ πως είναι πολύ σημαντικό να επιτύχουμε μια ισορροπία, έτσι ώστε και οι μικρότερες χώρες αλλά και οι μικρότεροι οργανισμοί να έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν στην χρηματοδότηση και σε αυτά τα προγράμματα. Ε, σίγουρα μεγάλοι όμιλοι, ε, ακαδημαϊκοί, ιδρύματα, πανεπιστήμια, σίγουρα ε, αυτά έχουν αριστεία και πρέπει να προωθούνται, όμως δεν πρέπει να παραμελούμε και τους μικρότερους. Διότι Πρέπει όλοι να έχουν ίσα δικαιώματα, ίσες ευκαιρίες και πρόσβαση. Πέραν αυτών, πιστεύω ότι και τα επιμέρους προγράμματα, αλλά και μεμονωμένοι πολίτες θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα συμμετοχής. Όχι μόνο μεγάλοι οργανισμοί, οι εκπαιδευτικά ιδρύματα, οι Βιομηχανική όμιλη. Θα ήθελα λοιπόν να ενισχυθεί η γνωμοδότηση σε αυτόν τον τομέα έτσι ώστε να είναι περισσότερο προσανατολισμένη προς το μέλλον και να δώσει προστιθέμενη αξία, να αυξήσει το βιωτικό επίπεδο των πολιτών. Σας ευχαριστώ πολύ. Και μετά την δική μου τοποθέτηση θα ήθελα να δώσω το λόγο στον, στην κυρία Τρούπελ, επόμενη σκιώδηση γήτρια. Θα, ευχαριστώ πολύ. Θα ξεκινήσω με ένα πολιτικό σχόλιο. Κατανοώ πως ε, εντοπίζεται μια ανισορροπία ανάμεσα σε, τα ανατολικά και τα δυτικά κράτη στη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, όμως με βάση αυτό το επιχείρημα θα σας πάω στην ε, Βουδαπέστη, στο Πανεπιστήμιο ε, που χρηματοδοτείται από τι Ηνωμένε Πολιτείε και απειλείται η ίδια του ύπαρξη αυτή τη στιγμή. Είναι ένα πανεπιστήμιο το οποίο δίνει έμφαση στην ε, φιλοσοφία, στις τέχνες, στον πολιτισμό. Χρειάζεται προσοχή, να μην, ε, παρα, να μην ε, παρα, γνωρίζουμε αυτό που γίνεται εκεί πέρα. Αυτό το εκπαιδευτικό ίδρυμα είναι πάρα πολύ σημαντικό για του νέου στην Ουγγαρία. Ναι, για μένα αυτό είναι σημαντικό. Εσεί έχετε την ευκαιρία να μιλήσετε, αφήστε και εμένα λοιπόν να το κάνω. Όταν καταφέρεστε εναντίον τη ε, Ευρώπη, όταν μιλάτε για ανισορροπίε, ε, να πρέπει να, να, πρέπει να αναγνωρίζουμε ότι ε, αυτό είναι αμφίδρομο. Και κάτι άλλο τώρα για τον ορίζοντα Ευρώπη. Νομίζω πως ως Επιτροπή Πολιτισμού είναι προς το συμφέρον μας να συνδέσουμε το πρόγραμμα Connecting Europe με τον ορίζοντα Ευρώπη. Ακριβώς διότι τα ο στόχος είναι ίδιος. Υπάρχει μία έκθεση στην Επιτροπή Ήτρε για τις ε, δημιουργικές βιομηχανίες και πολύ, για πολύ καιρό συζητούσαμε ε, αν θα έπρεπε να ασχοληθούμε με αυτό, αν είναι αρμοδιότητά μας. Όμως ο πολιτισμός είναι αρμοδιότητά μας και ε, πολύ σωστά αυτό. Δεν είναι βέβαια όλα ίδια, όμως ας δούμε τα, αυτά που μας ενώνουν, την ε, μόδα, την αρχιτεκτονική, όλες τις ε, δημιουργικές βιομηχανίες. Οφείλουμε να πείσουμε τους συναδέλφους μας ότι ο πολιτισμός ανήκει και εκείνο στις δημιουργικές βιομηχανίες, χωρίς να όμως να είναι το ίδιο και το αυτό. Εάν θέλουμε λοιπόν περισσότερη χρηματοδότηση πρέπει να το φροντίσουμε. Και ένα παράδειγμα, όταν ξεκίνησε η ψηφιακή επανάσταση στο Silicon Valley είδαμε το αποτέλεσμα. Είδαμε ότι η Apple είναι η πιο επιτυχημένη εταιρεία όλων των εποχών και, είδαμε, και γνωρίζουμε όλοι ότι ο Steve Jobs ξεκίνησε ως χίπης και έδωσε έμφαση στο σχεδιασμό και όλες οι συσκευές που δημιούργησε, το iPhone ας πούμε, είναι ένας συνδυασμός ε, σχεδιασμού και υψηλής τεχνολογίας. Αυτό είναι ένα άριστο παράδειγμα του ε, ότι κάτι τόσο ε, όμορφο και κομψό αισθητικά μπορεί να είναι και επιτυχημένο. Αυτό να το πάρουμε παράδειγμα και στην Ευρώπη. Δείτε ας πούμε τι γίνεται στη Γαλλία. Η βιομηχανία ειδών πολυτελείας της Γαλλίας έχει τα μεγαλύτερα κέρδη στην Κίνα. Αυτό μας δείχνει ότι οι δημιουργικές βιομηχανίες ανήκουν στον ορίζοντα Ευρώπη και συνδέονται στενά με τον πολιτισμό παρότι δεν είναι το ίδιο πράγμα. Γι' αυτό νομίζω θα πρέπει να υπερασπιστούμε τα συμφέροντά μας εκεί, χωρίς βέβαια να ε, παραμελούμε ότι χρειάζεται να υπάρχει και ένα ξεχωριστό πρόγραμμα στήριξης του πολιτισμού. Όμως πρέπει ο πολιτισμός να ανήκει στις δημιουργικές βιομηχανίες και να λαμβάνει την ε, αντίστοιχη στήριξη. Υπάρχει επίσης και χρηματοδότηση από διάφορα ταμεία, το Ταμείο Γιούγκερ για παράδειγμα, ε, ο πολιτισμός θα πρέπει να ανήκει σε αυτό, διότι είναι αναπόσπαστο κομμάτι της οικονομικής πολιτικής στην Ευρώπη, παρότι δεν είναι αμυγός οικονομικό, οικονομική, ε, οικονομικές διαστάσεις του. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Σόιντροβα έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Να προσθέσω κάτι μόνο Η κυρία Τροπελή, προηγούμενη ομιλήτρια, μίλησε για το θέμα της συνεργασίας και της σύνδεσης με το πρόγραμμα Creative Europe. Αυτό βεβαίως ε, είναι σωστό, αλλά μην ξεχνάμε και το Ταμείο Συνοχής. Η πολιτική συνοχή είναι εξαιρετικά σημαντική, ιδιαίτερα για τις νέες χώρες, για τα νέα κράτη-μέλη, διότι με αυτόν τον τρόπο χρηματοδοτούνται υποδομές για την καινοτομία και ακριβώς εκεί, σε αυτό το τομέα, θα πρέπει να δούμε τις αντιστοιχίες και τον συνδυασμό που μπορεί να γίνει. Είναι σημαντικό το Horizon Europe βεβαίως να συνδυαστεί και να είμαστε σαφείς στις προτεραιότητες που θέλουμε να θέσουμε. Η κυρία Ward. Νομίζω ότι βεβαίως υπάρχουν πολλοί συνδυασμοί μεταξύ αυτών των πρωτοβουλειών και άλλων, όπως παραδείγματο χάρη η ατζέντα στην καθώς και οι προτάσεις της Επιτροπής για συνδυασμό των ε, σπουδών που έχουν σχέση με τα επιστημονικά τους επιστημονικούς κλάδους, τους μηχανικούς, τα μαθηματικά και τον καλλιτεχνικό τομέα. Θα πρέπει να δούμε λιγάκι πιο γενικά τα προγράμματα αυτά και να δούμε τι είναι το καλύτερο για τους νέους της Ευρώπης, τι είναι καλύτερο για τα πανεπιστήμια μας, για τους ερευνητές, για την ερευνητική κοινότητα στην Ευρώπη που αντιμετωπίζουν σήμερα δυσκολίες αλλά και προκλήσεις. Και είναι σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε ότι ο πολιτισμός πρέπει να βρίσκεται σε όλα αυτά τα προγράμματα. Εγώ επί χρόνια ήμουν σε ένα πρόγραμμα για το συνδυασμό πολιτικής και επιστημονικού κλάδου. Και ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον το ότι πέρσι συνεργάστηκα με άτομα που προερχόταν από την κοινότητα των μεταναστών και η συνεργασία μας ήταν εξαιρετική. Με αυτόν τον τρόπο αποδεικνύουμε ότι πραγματικά εμείς μπορούμε να είμαστε πρωτοποριακοί στις, στα σχήματα που προτείνουμε και αυτή η δημιουργικότητα θα πρέπει να επεκταθεί και σε άλλα προγράμματα. Σαφώς λοιπόν και θα πρέπει να στηρίξουμε την ε, πολιτιστική συνιστόσα του προγράμματος Horizon 2020 και σίγουρα θα πρέπει να στοχεύσουμε τη στήριξη του Πανεπιστημίου ε, της Βουδαπέστης. Πάρα πολύ μεγάλη ανησυχία υπάρχει και εννοείται ότι οι ανησυχίες βασίζονται και στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι καθηγητές, οι πολίτες, οι εκπαιδευτικοί γενικότερα που συνεργάζονται με το πανεπιστήμιο αυτό, αλλά και όλη η ακαδημαϊκή κοινότητα, η εκπαιδευτική κοινότητα στην Ουγγαρία. Είναι ανησυχητικά αυτά τα φαινόμενα και θα πρέπει να στηρίξουμε για άλλη μια φορά την Ουγγρική εκπαιδευτική κοινότητα. Ευχαριστώ πολύ για τα σχόλιά σας. Το θέμα αυτό είναι δεύτερη φορά που το αναφέρετε. Θα προτείνω στους συναδέλφους το θέμα του Πανεπιστημίου της Βουδαπέστης βεβαίως μπορεί να είναι θέμα προς αλλά δεν νομίζω ότι μπορείτε να λέτε ότι αυτό το πανεπιστήμιο έχει κλείσει. Είναι ανοιχτό, λειτουργεί, υπάρχουν βεβαίως συζητήσεις οι οποίες συνεχίζονται. Παρόλα αυτά, δεν έχει κλείσει το Πανεπιστήμιο. Η συζήτηση συνεχίζεται και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να προτρέχουμε οι αποφάσεις δεν έχουν ληφθεί. Εν πάση περιπτώσει δεν είναι σωστό πριν ληφθούν οι αποφάσεις να συζητούμε το θέμα αυτό. Ας το κλείσουμε λοιπόν. Και θα δώσω τώρα το λόγο στην Επιτροπή. Θέλετε να πείτε κάτι για το Horizon 2020? Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τον, την εξαιρετική συνεισφορά του εισηγητή και των σκιωδών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταρχήν θα αναφερθεί στις συνέργειες, στο συμπληρωματικό χαρακτήρα μεταξύ των προγραμμάτων Horizon Europe και Creative Europe. Είναι σαφές ότι θα πρέπει να ενισχυθούν κάποιες πτυχές έτσι ώστε η δημιουργικότητα στην Ευρώπη και ο πολιτισμός να συμβαδίσουν. Πρέπει λοιπόν να παίξει εδώ ο πολιτισμός ένα σημαντικό ρόλο στην ενίσχυση της δημιουργικότητας, και όσον αφορά τη σημασία των λέξεων, εμείς στην Επιτροπή προτιμούμε να χρησιμοποιούμε τη λέξη κλάδι και όχι ο κλάδος, ο τομέας, με την έννοια ότι υπάρχουν πολλές δημιουργικές λύσεις που μπορεί να δοθούν, αλλά όχι μόνο από έναν τομέα, τον τομέα της βιομηχανίας ή της οικονομίας. Προτιμάμε λοιπόν να χρησιμοποιούμε τη λέξη κλάδι στον πληθυντικό, έτσι ώστε η δημιουργικότητα να ξεπεράσει την καθαρά εμπορική οικονομική διάσταση και να εξαπλωθεί σε όλους τους τομείς της δραστηριότητας. Θα δώσω και το λόγο σε λίγο για να συμπληρώσει αυτά που θα πω στην συνάδελφό μου, αναφερόμαστε στα σχόλιά σας που αφορούν το SSH. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι αυτό το θέμα δεν αντιμετωπίζεται μόνο με το Horizon Europe. Το τρίτο πιλωτικό πρόγραμμα Πρόκειται για ένα θέμα που σαφώς θα πρέπει να περιέχεται σε όλα τα προγράμματα, σε όλο το Horizon Europe. Και... Το τρίτο κλάστερ δεν περιορίζεται μόνο σε αυτό τον τομέα. Σε κάθε περίπτωση Οι τομείς των ανθρωπιστικών σπουδών και των κοινωνικών επιστημών, αλλά και η καινοτομία σε άλλους τομείς έρευνας. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε πιο ανοιχτοί και επιτρέψτε μου να σας πω ότι βεβαίως συνέργειες δεν σημαίνει ότι όλα θα πρέπει να συμβούν στο Horizon Europe, αλλά και αλλού. Και πολύ σωστά είπατε κάποιος από εσάς ότι θα πρέπει να δούμε την συμπληρωματικότητα και αυτό βεβαίως και όσον αφορά την χρηματοδότηση. Και το ίδιο ισχύει και για όλα αυτά που πρέπει να δημιουργήσουμε στα πλαίσια του προγράμματος που χρηματοδοτείται από το ESF, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, για να απλοποιήσουμε τις δυνατότητες συνεργασίας, συνέργειας, με περισσότερη αποτελεσματικότητα και πιο απλό τρόπο συμμετοχής για όλους όσους θέλουν να παίξουν κάποιο ρόλο σε αυτές τις συνεργασίες. Θα πρέπει επίσης να αποφύγουμε τον πολλαπλασιασμό των ε, παρεμβάσεων προτείνουμε επιπλέον ε, αν θέλετε συμμετοχές ιδιαίτερα στα καινούρια clusters εμείς θα προτιμούσαμε να δούμε πώς θα γινόταν κάποια από τα θέματα αυτά να ενσωματωθούν στις υπάρχουσες δομές και κλάστερ. Αυτό εν μέρη συμβαίνει ήδη στους δημιουργικούς τομείς, στις αν θέλετε, πρωτοβουλίες όπως ε, για την πολιτιστική κληρονομιά. Βέβαια, μπορούμε να βελτιώσουμε την συμμετοχή, την αποτελεσματικότητα, αλλά ας μην πολλαπλασιάσουμε τις δυνατότητες συμμετοχής έτσι ώστε στο τέλος να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον εξαιρετικά περίπλοκο και πολύ δύσκολο ε, για όλους αυτούς που θέλουν να δραστηριοποιηθούν να το κατανοήσουν. Το STEAM, η ατζέντα, δεν αναφέρεται ουσιαστικά στο δεύτερο πυλώνα, αλλά στη βάση αυτού του πυλώνα που ουσιαστικά έχει σαν σκοπό την ε, συμμετοχή στην αριστεία αλλά και τη διεύρυνση όλων αυτών των δεξιοτήτων με σκοπό να συνεχίσουμε τη στήριξη που σήμερα υπάρχει στο Horizon 2020 για το STEAM και βεβαίως με στόχο την συμμετοχή νέων φοιτητών και μαθητών. Δεν θα αναφερθώ καθόλου στον προϋπολογισμό, σημειώνουμε αυτά που αναφέρατε, δεν έχω αρμοδιότητα να αντιδράσω για θέματα δημοσιονομικά. Και ολοκληρώνω τις παρατηρήσεις μου, εγώ τουλάχιστον, σε αυτό που πολύ σωστά είπατε όσον αφορά τα ανώτατα ακαδημαϊκά ευρωπαϊκά ιδρύματα, προτιμούμε να χρησιμοποιούμε ακαδημαϊκά ιδρύματα παρά τον όρο πανεπιστήμια. Συμφωνούμε με την έννοια των πανεπιστημίων, αλλά ξέρετε ότι υπάρχει και μια ιδιαίτερη πρωτοβουλία για την δημιουργία ενός δικτύου των Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων. Εσείς προτείνετε κάτι πιο ευρύ, πέρα δηλαδή από το δίκτυο για τα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια. Και γι' αυτό και θέλουμε να ακολουθήσουμε την πρότασή σας, αν κατανοώ αυτό που λέτε. Προτιμούμε λοιπόν να μιλάμε για ανώτερα, ανώτατα συγγνώμη, ε, ακαδημαϊκά ιδρύματα. Και όχι πανεπιστήμια μόνο. Ευχαριστώ πολύ. Αυτά. Σας ευχαριστώ πολύ, λέει η Πρόεδρος. Και θα ξαναδώσω το λόγο στον κύριο Μοργάνο για τρία λεπτά. Καταρχήν, σας ευχαριστώ Ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους ε, που πήραν το λόγο. Σημείωσα τις παρατηρήσεις σας και φυσικά θα τα συμπεριλάβουμε αυτά στις ε, τροπολογίες. Τώρα τόσο επί κομισιών μου φαίνονται σημαντικά. Εδώ θα πρέπει να συνεννοηθούμε. Νομίζω ότι ήταν ξεκάθαρη η σημερινή συζήτηση, δηλαδή η απέτηση να μπορέσουμε να έχουμε μεσοπρόθεσμα τη δυνατότητα ενός ελέγχου μιας επαλήθευσης για το τι γίνεται. Αν δεν προβλέπεται ο έλεγχος αυτός, αυτή η επαλήθευση, τότε γίνεται πιο πολύπλοκο και από την πλευρά του Κοινοβουλίου να υλοποιήσει τα καθήκοντά του στην περίπτωση αυτή και η Επιτροπή να μπορέσει να επαληθεύσει αν σε επίπεδο Επιτροπής ακολουθούνται οι πολιτικές κατευθύνσεις του Κοινοβουλίου. Τώρα, σε σχέση με την ορολογία και αυτό είναι σχετικό. Τι σημαίνει σήμερα τομέας. Κλάδος είναι ένας πολύ ευρύς όρος. Δηλαδή από τη στιγμή που χρησιμοποιώ ένα τέτοιο ευρύ όρο ε, δεν μπορώ να επαληθεύσω τι συμβαίνει στα προγράμματα. Δηλαδή, ή θα συνεννοηθούμε για το τι θέλουμε να πούμε, γιατί όταν ε, μιλώ για πολιτιστική και δημιουργική βιομηχανία, αυτό είναι κάτι ξεκάθαρο. Ο όρος είναι ε, το industry, βιομηχανίας πολιτισμού και της δημιουργίας. Έτσι λοιπόν, Α, το ένα είναι να βρούμε έναν τρόπο που να μπορεί να ανοίγει και όχι να κλείνει τις δυνατοιτές μας και τη στιγμή που μιλάμε για ανώτατα εκπαιδευτικά οδρήματα, ε, το θέμα είναι η άλλη κατάρτιση που θα μπει δηλαδή οι ερευνητές που στη συνέχεια ε, μπαίνουν στα ακαδημαϊκά ιδρύματα ή προσπαθούν ε, να μπουν, ε, παραδείγματο χάρη, σε κάποια ακαδημαϊκά ε, ιδρύματα και στη συνέχεια πηγαίνουν σε επιχειρήσεις για να εφαρμόσουν την ερευνά τους. Εγώ τον όρο πανεπιστήμιο δεν μπορώ να τον ξεπεράσω. Ίσως θα πρέπει να κάνουμε ένα κατάλογο για να είναι ξεκάθαρα τα πράγματα ή διαφορετικά, επιτρέψτε μου την εντύπωση που έχω, Δηλαδή εδώ υπάρχει κάτι ε, που είναι ε, υπερβολικά προσδιόριστο και δεν επιτρέπει στο Κοινοβούλιο να ελοπίσει τα καθήκοντά του, δηλαδή είτε το καθήκον αξιολόγησης είτε επαλήθευσης των συνεργειών. Γιατί, όπως ε, είπαμε πριν, το ένα είναι να δούμε ποια είναι τα εργαλεία που χρησιμοποιούμε με τις κατάλληλες συνέπειες. Φυσικά το πνεύμα είναι μεγίστη συνεργασίας. Όμως, νομίζω είναι σημαντικό για όλους να μπορέσουμε να λάβουμε υπόψη αυτές τις δύο πτυχές που είναι απολύτως σχετικές. Και επιτρέψτε μου να το πω, ακόμη και η τεχνική χρόνη είναι πραγματικά πάρα πολύ στενή. Και θα ήθελα να ευχηθώ να μην επαναληφθεί. Γιατί δεν επιτρέπει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να υλοποιήσει τα καθήκοντά του εις βάθος. Και αυτό το θέμα δεν είναι μόνο πολιτικό, αλλά είναι πάρα πολύ σχετικό. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Μπορούμε να ολοκληρώσουμε λοιπόν το σημείο αυτό. Η προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών είναι 10 Σεπτεμβρίου, όχι 5 Σεπτεμβρίου λέει η Πρόεδρος, στις 2 το μεσημέρι. Και τώρα προχωρούμε στο επόμενο θέμα της ημερησίας διάταξης ειδικέ διατάξεις ε, για το στόχο Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασίας, Interreg, με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και των Μηχανισμών Εξωτερική Χρηματοδότησης. Η συγγήτρια είναι η Μαρλέν Μίτσι. Προθεσμία κατάθεσης των τροπολογιών είναι η 10 Σεπτεμβρίου στις 5 το απόγευμα. Η Επιτροπή Πολιτισμού θα ψηφίσει στις 10 Οκτωβρίου και η αρμόδια επιτροπή, η Ρέτζη, στις 21 Νοεμβρίου. Και καθώς η κυρία Μίτσι δεν είναι εδώ, ο κύριος Μοργάνο θα ξαναπάρει το λόγο και θα μας ε, παρουσιάσει την εκθέση αυτή εξ ονόματος ε, της κυρίας Μίτση. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, προφανώς εγώ θα διαβάσω το κείμενο της ε, συναδέλφου της κυρίας Μίτση Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα καταρχήν να εκφράσω ε, την λύπη μου που δεν μπορώ να είμαι παρούσα σήμερα. Θα σας ε, παρουσιάσω υπό αυτό το σημείο τους, ε, τα κυρία σημεία των τροπολογιών που περιέχονται στην πρόταση γνωμοδότησης σχετικά με τον κανονισμό ε, που αφορά το πρόγραμμα Interreg 2021-2027 ε, σε σχέση με τις ε, ειδικέ διατάξεις για το στόχο Ευρωπαϊκή Δευκή Συνεργασία που υποστηρίζεται και από το ΕΤΠΑ και τους μηχανισμούς εξωτερικής χρηματοδότησης. Σύμφωνα και με το πνεύμα του Ευρωπαϊκού Έτους Πολιτιστικής Κληρονομιάς, οι τροπολογίες που προτείνονται στην γνωμοδότηση της συναδέλφου Μίτση θέλουν να εγγυθούν ε, μια μεγαλύτερη ελεπίδραση μεταξύ αυτού του προγράμματος ε, και ε, των, πολιτικών στον τομέα του πολιτισμού, της παιδείας, του αθλητισμού και της νεολαίας. ή τροπολογίες που συμπεριλαμβάνονται στη γνωμοδότηση που θα στελεί στην Επιτροπή Ρέτζι εισάγουν με σαφήνεια την πολιτιστική και εκπαιδευτική διάσταση της διασυνοριακής συνεργασίας που προβλέπεται στο πρόγραμμα Interreg είτε μεταξύ των περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε μεταξύ αυτών και περιφερειών μη Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, η ε, παιδί, ο πολιτισμός αλλά και ο αθλητισμός και οι πολιτικές για την ΛΕΕ είναι απαραίτητες πτυχές της οικονομικής και κοινωνική ανάπτυξη και της πρόθεση της εδαφική συνοχής προκειμένου να αμβληθούν ε, οι παρεξηγήσει και τα γλωσσικά εμπόδια και προκειμένου να προωθηθεί μια αποτελεσματική συνεργασία. Εκτιμώ ιδιαίτερα το που αναφέρεται ε, στην ενίσχυση των ικανοτήτων μέσω των θεματικών ε, πλατφόρμων της Smart Specialization ε, μαζί με ε, έναν εξυγχρονισμό στον τομέα της βιομηχανίας, της γεωργίας και της ενέργειας. Αυτά αποτελούν ε, ενάρετα παραδείγματα που έχουν αναπτυχθεί πρόσφατα, όπως παραδείγματος χάρη με το δίκτυο RIC που αφορά ε, την Περιφερειακή Πρωτοβουλία για τον Πολιτισμό και τη Δημιουργικότητα και έχει ως στόχο να συνδέσει ε, τα διάφορα κράτη-μέλη που έχουν ξεκάθαρο όραμα επί των πολιτικών αυτών. Έτσι, λοιπόν, ε, είναι προτεραιότητα να έχει περισσότερο κεντρικό ρόλο αυτό στην προγραμματική περίοδο 2021-2027. Ε, αυτό το σχέδιο συμβαδίζει με τους στρατηγικούς στόχους ε, της νέας πολιτικής 2027 που θέλει μια Ευρώπη πιο κοινωνική και πιο κοντά στους πολίτες. Ε, θέλω να υπογραμμίσω λοιπόν ότι το Ίντερεκ θα πρέπει να κάνει ομαδικό παιχνίδι με τα λοιπά προγράμματα και να προβλέψει ενάρετη λιλεπίδραση. Επομένως, ορθά τονίζουμε την πρόσβαση στην ε, εκπαίδευση και ε, στον πολιτισμό ε, σε διεθνικό επίπεδο, την αύξηση της κινητικότητας των νέων και την πρόθεση της κινητικότητας των καλλιτεχνών. Αυτά αποτελούν καινοτομίες του προγράμματος και συμπεριλαμβάνονται στην πρόταση γνωμοδότησης. Έτσι λοιπόν, εξ ονόματος συναδέλφου Μίτση, ζητώ να υποστηρίξετε τις τροπολογίες που προτείνονται και ενδεχομένως τις επόμενες μέρες να παρουσιάσετε καινούριε, λαμβάνοντας υπόψη και την προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών. Ευχαριστώ πολύ. Δεν έχουν ορίσει ακόμα όλες οι πολιτικές ομάδες και οι συγητή. Οι σκιώδεις συγητές δεν είναι όλοι παρόντες. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα σε αυτό το σημείο να ε, ζητήσω από όποιον θέλει να πάρει το λόγο. Εάν δεν θέλει καλή το λόγο, τότε θα δώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τυχόν σχόλια. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Μοργάνο για την παρουσίαση των τροπολογιών της, ε, που προτείνει η κυρία Μίτση. Θα ήθελα και εγώ να πω δύο λόγια, διότι θεωρούμε ότι οι τροπολογίες ασχολούνται με πολύ σημαντικά θέματα και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είναι κατά αυτών των προτάσεων επί της ουσίας. Θεωρούμε πως είναι όντως πολύ σημαντικό να υπάρξει ευαισθητοποίηση για πολλά θέματα στον τομέα της ε, εκπαίδευσης και του πολιτισμού που εμποδίζουν την ανάπτυξη περιφερειών που συμμετέχουν στους στόχους της Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας. Αυτό είναι και ο λόγος που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει συγκεκριμένο κανονισμό για την ε, εδαφική συνεργασία. Αυτά τα πολύ συγκεκριμένα θέματα που τονίζονται εδώ σε πολλές περιπτώσεις αφορούν τον σχεδιασμό. Τονίζονται αρκετά στοιχεία από αυτά και είναι πολύ σημαντικό να διευκρινιστεί ο γενικότερος στόχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έτσι ώστε να μειωθεί σε έκταση το κείμενο και να εστιάσει στα ουσιώδη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί πως στον, στο παρόν σχέδιο περιλαμβάνονται πολλές από αυτές τις προτάσεις. Δεν διαφωνούμε δηλαδή επί της ουσίας, αλλά δεν θεωρούμε πως ε, σε αυτό το στάδιο είναι σημαντικό να ε, συμπεριληφθούν, ακριβώς γιατί καλύπτονται από το αρχικό, την αρχική, από το αρχικό σχέδιο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ήθελε δηλαδή μία μινιμαλιστική προσέγγιση στο κείμενο, ακριβώς διότι η εμπειρία μας δείχνει ότι ε, το εφιστάμενο πλαίσιο παρέχει ασφαλεία δικαίου στους ε, διάφορους φορείς και θα θέλαμε λοιπόν ο σχεδιασμός να παραμείνει λιτός. Να τονίσω ένα στοιχείο που αφορά τους δύο συγκεκριμένους στόχους που Υπάρχει πρόταση να προσθεθούν. Ο έχει να κάνει με την εκπαίδευση και την αμοιβαία αναγνώριση πιστοποιητικών, διπλωμάτων και άλλων τίτλων κατάρτισης και ο άλλος αφορά την πολιτισμική κληρονομιά. Θεωρούμε πως ε, και σε αυτόν τον τομέα έχουμε ήδη καλύψει τα ζητούμενα, ακριβώς γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικός. Και αναφέρομαι στο σημείο Β. Και εδώ νομίζω πως όσον αφορά την αμοιβή αναγνώριση διπλωμάτων ε, έχουμε καλύψει και αυτόν τον στόχο το, όσο και τα υπόλοιπα θέματα που αναφέρονται στην ε, τροπολογία 10. Θεωρούμε πως ε, τόσο στον κανονισμό για ταμεία συνεχής όσο και σε εκείνον το Ταμείο περιφερειακή Ανάπτυξης συμπεριλαμβάνονται αυτά τα στοιχεία. Τα καλύπτουν λοιπόν και δεν θεωρούμε απόλυτα αναγκαίο να ε, υπάρχουν αυτές οι δύο τροπολογίες. Είναι τεχνικού χαρακτήρα αυτές οι διευκρινήσεις, όμως θέλουμε να κρατήσουμε το κείμενο λιτό. Γι' αυτό κάνουμε αυτή την παρατήρηση. Και ε, κλείνοντας θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους για την ε, δουλειά σας, τη γνωμοδότηση αυτή. Ευχαριστώ πολύ. Και σε αυτό το σημείο νομίζω ότι μπορούμε να ολοκληρώσουμε και αυτό το κομμάτι. Να σας ενημερώσω ότι η επόμενη συνεδρίαση θα λάβει χώρα στις 24 Σεπτεμβρίου από τις 2.30 έως τις 6.30 το απόγευμα. Θα ήθελα λοιπόν να παρακαλέσω τους συναδέλφους να λάβουν υπόψη ότι στις 24 Σεπτεμβρίου θα ξεκινήσουμε μισή ώρα νωρίτερα. Σας ευχαριστώ πολύ για τη συμμετοχή σας, ευχαριστώ πολύ και τους διερμηνείς και σας εύχομαι καλό βράδυ.